Dear colleagues, συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και τον Επίτροπο στις 11. Ξεκινάμε αμέσως με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται, χωρίς αλλαγές. Για το επόμενο θέμα, ανακοινώσεις του Προέδρου να σας πω πως η συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τις 19 ε, Μαρτίου αναβάλλεται. Ανταυτού θα έχουμε την 3η 31 Μαρτίου μια συνεδρίαση μισής μέρας το απόγευμα. Θα σας στείλουμε με email το νέο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες και ο συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών ε, της ε, συνεδρίασης της 27ης Ιανουαρίου εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει ε, μέχρι το τέλο της συνεδρίαση. τα πρακτικά θεωρείται ότι εγκρίνονται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ε, ρήπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους ε, μονάδες καύσης. Εισηγητή ο συνάδελφο, ο κύριος Ζήμπα και του δίνω αμέσως τον λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να πω πως ε, η πρόταση αυτή της ε, Κομισιόν σχετίζεται με το πρόγραμμα για το περιβάλλον μέχρι το 2020 το οποίο έχει ως σύνθημα να ζούμε εντός των ορίων του πλανήτη μας. Στόχο δημιουργία καλύτερης ποιότητας αέρα στην, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε γύρω στις 150.000 ε, μονάδες καύσης μεσαίου μεγέθους ε, με θερμική απόδοση μεταξύ 1 και 50 ΜΒ χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και θέρμανση κατοικιών, αλλά και στην βιομηχανία. Οι μονάδες αυτές λοιπόν εκπέμπουν επίσης διοξίδιο του θείου, του αζότου, καθώς και μικροσωματίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχουμε νομοθεσία για τις μικρές μονάδες καύσης κάτω του 1 ΜΒ. Είναι η οδηγία 2009 κάθετος 125 περί οικολογικού σχεδιασμού. Επίσης καλύπτονται και οι μεγάλες μονάδες καύσης. αποκαλύπτονται από την Αδικία 2010 75 περί βιομηχανικών εκπομπών. Οπότε η ρήπη από μεσαίου μεγέθους ε, μονάδες ε, δεν καλύπτονται συνήθως στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε η Κομισιόν εδώ πέρα εντόπισε ένα κενό στην ε, νομοθεσία. η πρόταση της Κομισιόν 0442 του 2013 έχει κάποιες προτάσεις για τη μείωση της ρήπανσης, ειδικά όσον αφορά τα οξύδια του αζότου, διοξίδιο του θείου και σωματίδια. Αυτό γίνεται μέσω του καθορισμού οριακών τιμών για, τα νέα, για τις νέες και τις υφιστάμενες μονάδες. Όλα αυτά ε, σχετίζονται και με την καταγραφή των μονάδων αυτών. Μια καταγραφή η οποία θα γίνει από τις εθνικές αρχές ε, με την μεταφορά αυτής της ε, νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα λοιπόν με την ιδέα αυτή περί καλύτερης ε, ρύθμισης ε, σκοπεύουμε εδώ πέρα να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και την υπερβολική γραφειοκρατία διατηρώντας άθικτους ε, τους ε, στόχους της αθικής ε, νομοθετικής πρότασης. Είναι λοιπόν φιλόδοξη η στόχη, εγώ θα ήθελα να τους κάνω λίγο πιο φιλικούς προς τις επιχειρήσεις, γιατί θα επηρεαστούν έτσι περισσότερο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και πολλές δημοτικές επιχειρήσεις. Επίσης, καλύπτονται και κάποια κτίρια κατοικίας σε κάποιες χώρες, π.χ. πολυκατοικίες, στις οποίες υπάρχει μια διαχείριση από τους ε, ενίκους, ε, οι οποίοι μπορεί επίσης να έχουν μια τέτοια μονάδα καύσης ε, μεσαιομογέθους και αυτοί καλύπτονται. Οι αλλαγές αυτές λοιπόν έχουν στόχο να γίνει πιο ρεαλιστική η εφαρμογή της οδηγίας για να βελτιωθεί όντως ε, η ποιότητα του αέρα. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά ε, αυτούς ε, που έχουν αυτές τις μονάδες ή την κοινωνία την ίδια. Γιατί όπως είπα, κάποιες από τις νέες αυτές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν ε, και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Τώρα, για να έρθουμε στην έκθεσή μου. Προτείνω να αλλάξουμε το άρθρο 2 για να εφαρμόσουμε το, για να προσαρμόσουμε το πεδίο εφαρμογής, με συγχωρείτε, και να δούμε το τι ρυθμίζεται ήδη. Παραδείγματος χάρη από την οδηγία περί βιομηχανικών ρήπων την 2975 του 2009 και άλλα νομοθετήματα. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρχουν περιτά βάρη στις ε, εταιρείε ε, και στους ιδιώτε που έχουν τέτοιε μονάδε Αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά τη διάρκεια της ε, διαβούλευση ε, με ρώτησαν αρκετέ φορές το εάν το κόστο, μείωση των εκπομπών δικαιολογείται. Οπότε είναι σημαντική η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος και τα έχω συμπεριλάβει αυτά στο παράρτημα 2 και πρέπει όπως είπα να υπάρξει μια κατάταξη με βάση την θερμική απόδοση των μονάδων. Ε, ένα μέχρι 5 ΜΒ, 5 με 15 και μετά 15 με 50 για να μην υπάρξουν ε, παρερμηνίες ε, και ασάφειες. Ε, για τον λόγο αυτό πρότεινα και κάποιες αλλαγές στο άρθρο 5. Τώρα να αναφερθώ στα άλλα ζητήματα τα οποία είναι ακόμη εκκρεμή γιατί η διαδικασία διαβούλευσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν έχω ακόμα συμπεριλάβει όλες ε, τις ε, τροπολογίες. Ε, κάποιες από αυτές ήρθαν μετά την προθεσμία. Οπότε υπάρχουν κάποια ζητήματα Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, η εκχώρηση δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένες ε, λύσεις. Το δεύτερο βεβαίω είναι ένα ζήτημα του πώς γίνεται η αναφορά και κατά την άποψή μου όποια οποιαδήποτε νέα πρόταση και ρύθμιση που αφορά το περιβάλλον και όχι μόνο επιβάλλει σε επιχειρήσεις μια υποχρέωση να αναφέρουν στις αρχές το τι κάνουν και αυτή συχνά περιλαμβάνει τα ίδια δεδομένα τα οποία τα στέλνουν πολλές φορές σε διαφορετικά θεσμικά όργανα που έχουν διαφορετικές ε, βάσεις δεδομένων. Αν υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση λοιπόν προτείνω ναι, υπάρχει κάποιο έλεγχο, αλλά δεν νομίζω πω αυτή είναι η ιδανική λύση. Είτε για την Κομισιόν, είτε για τα κράτη-μέλη. Συχνά λοιπόν. Και η αναφορά αυτών των διοικητικών δεδομένων είναι αρκετά μεγάλο βάρος και αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τις αναφορές αυτές για να γίνονται από κοινού με πράγματα τα οποία προβλέπουν άλλοι κανονισμοί. Οι ειδικοί όμως μου είπαν πως δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν κάτι τέτοιο. Τώρα θα μπορούμε να τα αφήσουμε ανοιχτό το ζήτημα προς στιγμή και να δούμε τους, ε, την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών και να δούμε αν υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς έτσι ώστε όλες ε, οι αναφορές να στέλνονται σε έναν φορέα και να διευκολυνθούν κάπως ε, οι επιχειρήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε ήταν η σχέση μεταξύ μείωσης κάποιων εκπομπών και η αποτελεσματικότητα των ε, μονάδων αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Δεν έχουμε μελέτες που να μας δίνουν μια πραγματική εικόνα του εάν οι αυξημένες εκπομπές ε, επηρεάζουν ε, την αποτελεσματικότητα παραγωγής ενέργειας και αν Άρα η μείωση των εκπομπών θα οδηγήσει συνολική μείωση των, των ρήπων, θα μειώσει συνολική μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Κάτι άλλο που προέκυψε κατά την σύνταξη της έκθεσης είναι το θέμα των ε, πήγων ε, μικροσωματιδίων. Η πρόταση της ε, Κομισιόν μιλάει για πηγές οι οποίες ε, λειτουργούν τουλάχιστον 500 ώρες ε, το χρόνο και λέει πως θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή του Συμβουλίου και να αυξηθεί το νούμερο αυτό στις χίλιες ώρες το έτος. Και μάλιστα να είναι ένας μέσος όρος ε, πέντε ετών οι ώρες αυτές. Αυτό είναι δύσκολο γιατί πραγματικά επηρεάζει τις χώρες ε, στη Βόρεια Ευρώπη όπου είναι οι χειμώνες πιο δύσκολοι και 500 ώρες λειτουργίας για μέσες ε, μονάδες δεν επαρκούν δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν. Και μου είπαν ότι έχουν αυτές τις ανάγκες. Νομίζω ότι καταφέραμε νομίζω να βρούμε μια θετική λύση για τις μονάδες καύσης οι οποίες είναι σε νησιά ή σε ενεργειακά όπως λέμε νησιά π.χ. τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάποιες στο βορρά. Συντάσσοντας λοιπόν την έκθεση αυτή έπρεπε να κάνω και μία επιλογή. Καθώς έχουμε φαινός την ε, αποτελεσματικότητα της ε, παραγωγής ενέργειας και την στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την άλλη έχουμε την εκπομπή μικροσωματιδίων. Αυτό αφορά επίσης και τις βορείς χώρες ε, που χρησιμοποιούν ε, το ξύλο ως καύσιμο. Τον ε, προσαρμόσουμε λοιπόν τις μονάδες αυτές τους νέους κανονισμούς θα κόστιζε περισσότερο από την επένδυση που έχει γίνει στις ίδιες τις μονάδες, από όσο κοστίζουν οι ίδιες οι μονάδες. κανόνες για λέβητες ε, βιομάζας είναι επίσης ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ήθελα να πω πως ε, ελπίζω πραγματικά να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Οι αρχικές επαφές με τους σκιώδεις εισηγητές ήταν πολύ θετικές. Εγώ ε, να δεχτώ οποιοδήποτε επιχείρημα έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Είμαι ανοιχτό. σε σχέση με την έκθεση αυτή και θα προσπαθήσω να δράσω με έναν τρόπο που θα είναι προς το συμφέρον της έκθεσης για να ψηφιστεί τελικά. Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τον πρώτο κύκλο τοποθετήσεων με τους κοιόδης ηγητές. Παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι σχετικά, έτσι ώστε στις 11 να έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ο κύριος Παολούτσι. Grazie Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ε, το οποίο καλύπτει ένα αριθμιστικό κενό, που όπως παρατηρήσαμε αφορά ε, πολλές χιλιάδες επιχειρήσεων. Είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, οπότε δεν θα σταθώ στη σοβαρότητα των στοιχείων περί ρήπανσης. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η ρήπανση αποτελεί το βασικό αίτιο για την προορυθμισιμότητα, ε, επίσης ε, γνωρίζουμε ε, πόσο σοβαρές, σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι το κόστος που πληρώνουν τα εθνικά μας συστήματα υγείας για τις ασθένειες που απορρέουν από την ρήπανση. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν μινιμαλιστική προσέγγιση ή να υποτιμούμε το θέμα όταν συζητάμε πώς θα βελτιώσουμε την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα. Δεν θέλουμε να καταστήσουμε δύσκολη τη ζωή των επιχειρήσεών μας. Γνωρίζουμε ότι η ευρωπαικη επιτροπη σιγουρα δεν θελουμε να καταστησουμε δυσκολη τη ζωη των επιχειρησεων μας γνωριζουμε οτι ρήπανση ατμοσφαιρική δεν εξαρτάται μόνο από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από την θέρμανση του πλανήτη αλλά και από την κίνηση και γνωρίζουμε ε, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει και τις δύο αυτές πηγές ρήπανσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση είναι λογική αλλά δεν συμφωνώ ε, να καταστήσουμε απόλυτα δεσμευτική αυτή τη δέσμευση, αυτή την, ε, αυτό το, κανονισμό. Πιστεύω πως η πρόταση Κομισιόν είναι θαραλέα και αποτελεί το αντίβαρο σε ορισμένες προτάσεις σε ανατολισμού του Συμβουλίου που κατά τη γνώμη μου αποδυναμώνουν ή ακόμα και ε, εκφυλίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Για να τα πω ξεκάθαρα και ειλικρινά, οι θέσει του Συμβουλίου δεν θεωρώ πως είναι βάση για να φτάσουμε σε μια αποδεκτή συμβιβαστική λύση. Α πούμε τώρα στην ουσία διάσταση των εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να σκεφτούμε χωρίς καμία προκατάληψη όσον αφορά ε, τις διαστάσεις και τις διαβαθμίσεις των μέτρων. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και εγκαταστάσεις 1 με 5 ΜΒ που αποτελούν ε, ε, μέχρι το 20% των εμπορευμάτων, της παραγωγής εμπορευμάτων, είναι υπεύθυνα για το 35% της ρήπανσης. Επί της ουσίας, η επιλογή ενός ε, καθεστώτος ε, καταγραφής, ορισμένα κρατημέλη έχουν ε, τέτοιο σύστημα ήδη όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Πολύ αυστηρό μάλιστα σύστημα. Θα ήταν λάθος το να ακυρώσουμε όλη τη δουλειά αυτή που έχει γίνει και άρα λοιπόν είναι προσδεκτή η ιδέα να αφήσουμε στα κρατη τη διαδικασία συστήματος αδειοδότησης καθώς και καταγραφής μητρώου των εργοστασίων. Τώρα, εγώ θα περιοριστώ στο να, στο να παρατηρήσω ότι συμμερίζομαι την προσέγγιση που διάβασα ε, στην Ήτρε, σύμφωνα με την οποία η κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να υπόκειται σε διπλή ρυθμίσει. Ο ορισμός ε, η φυστάμενη συγκατάσταση νέα εγκατάσταση. Κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερη η πρόταση που έχει προτείνει αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα η Κομισιόν. Γιατί έτσι θα πρέπει επίση να απλοποιήσουμε τον κατάλογο των κυρώσεων που προτείνονται. Πάντα επί της ουσίας όσον αφορά το χρόνο, την προθεσμία για την καταγραφή, την διαδότηση των εγκαταστάσεων. 2025, 10 χρόνια από τώρα για τα εγκαταστάσεις πάνω από 5 ΜΒ και 2003, δηλαδή 15 χρόνια από σήμερα, είναι τα εργοστάσια πάνω από τα 5 ΜΒ. Πιστεύω πως ε, δεν είναι επαρκή σε αυτή η πρόταση, είναι αδύναμη. Η Κομισιόν βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο καταγραφής ε, προτείνει μόνο 13 μήνες, ε, όχι 15 χρόνια. Εγώ πιστεύω πως δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή την πρόταση των 13 μηνών. Τώρα, παράδειγμα 2. Έχουμε τρει διαφορετικέ θέσει. Σύμφωνα με την Κομισιόν θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί από το 2025 μέχρι το 2030, ανάλογα με το αν ε, τα εργοστάσια είναι απόδοσης πάνω από 5 ε, ΜΒ ή κάτω από 5 ΜΒ. Μετά, διάκριση ανάμεσα στις διάφορες διαβαθμίσεις ε, μεγέθους. 1 ε, με 5, 5 με 15, 15 με 50 ΜΒ. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να περιορίσουμε ε, διαφορετικά από την οδηγία του 75 που είχε ορίσει τα εργοστάσια μέχρι 50 ΜΒ. Πρέπει ωστόσο να περιορίσουμε τις εξαιρέσεις και να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα μέγιστο όριο. Παράρτημα 3 που ορίζει τη όρια όσον αφορά ε, την οδηγία 2008. Κατανοώ ότι η ρήπανση η ατμοσφαιρική δεν εξαρτάται μόνο από τις βιομηχανικές εκπομπές, αλλά θα ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου να καταργηθεί το παράρτημα 3. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια ενώπιον τη σοβαρότητα της κατάστασης σε ορισμένες περιοχές των πόλεων μας και των χωρών μας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά θα υπογραμμίσω μόνο κάποια και θα προσπαθήσω να κλείσω γρήγορα θα πρέπει να εμβαθύνουμε βέβαια σε όλα αυτά οι περιοχές, τα νησιά που είναι υπερπεριφερειακές και είναι απομονωμένες, το θέμα της βιομάζας, τα εργοστάσια που λειτουργούν για συγκεκριμένες ώρες και τα δημόσια μέτρα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Προτάσεις στις οποίες θα πρέπει να βρούμε κοινές, κοινά στοιχεία. Έπειτα, ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόταση της Κομισιόν ε, για να μην υπάρξουν παραθυράκια. Να δώσω το παράδειγμα των των εργοστασίων που σωρεύουν διάφορα, διάφορες εκπομπές ε, καθώς και για τις ε, συστάδες ή ομίλους εργοστασίων ή ε, εργοστασιακές ζώνες. Να δούμε επίσης και ποιες είναι οι εκπομπές στη διάρκεια ζωής των εργοστασίων. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Ουισνιέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Ξιμπ για την ε, έκθεση αυτή. Η συζήτηση ξεκίνησε το Δεκέμβριο. Τότε μιλήσαμε για το σημαντικό θέμα της αναλογικότητας του κόστους το οποίο απορρέει από αυτούς τους κανόνες και βαρύνει επιχειρήσεις ε, και ιδιώτες. Το θέμα της αναλογικότητας έχει τρεις πτυχές. Πρώτον, να το ξεχωρίζουμε μεταξύ διαφορετικών ε, ισχύων, ε, το ότι δεν έχουμε ιδιαίτερους κανόνες για περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα οικολογικού περιεχομένου και χαίρομαι που ο εισηγητής προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της αναλογικότητας ε, της ε, πρότασης της ε, Κομισιόν. Είναι σημαντικό να χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες, ένας 5, 5, 15, 15, 50 ΜΒ. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε διάκριση σε ό,τι αφορά τους κανόνες που ε, τους ε, επιβάλλονται σε κάθε εγκατάσταση. Ε, οι μικρότερες εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, έχουν, πρέπει να έχουν πιο απλούς και λιγότερο επιβαρυντικούς κανόνες, διότι μολύνουν λιγότερο. Η σχέση κόστους-οφέλους επίσης είναι διαφορετική για κάθε μία από τις κατηγορίες. Οπότε υποστηρίζω τον εισηγητή. Ε, επίσης είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ νομοθετικών κειμένων, όπως λέει ο εισηγητής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται, ίσως θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο μακριά από αυτό που λέει ο εισηγητής. Αυτοί οι κανόνες, αυτά τα πρότυπα, ίσως δεν θα πρέπει να είναι, δεν θα πρέπει να είναι ε, υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει το κράτος μέλος. Αυτό το δέχομαι ως ιδέα. Τα κράτη-μέλη ενδεχομένως θα μπορούν να επιβάλλουν ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες, αν το επιθυμούν. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην ε, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τα ελάχιστα. Θέλουμε να ε, σταθμίσουμε πολύ σωστά τα μέτρα που θα πάρουμε, διότι μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικά, σημαντικό υψηλό κόστος επί των επιχειρήσεων. Οι εγκαταστάσεις ε, κάψης μεσαίου μεγέθους είναι πολλές φορές καυστήρες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας σε πολύ μικρή κλίμακα. Οι μισοί καταναλωτές στην χώρα μου χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μονάδες καύσης. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Βέβαια η τηλεθέρμανση μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό ε, ζήτημα, αλλά για μας είναι. Επίσης ε, χρειάζεται ε, ανανέωση του εξοπλισμού, διότι χάνουμε πολλή ενέργεια. Όμως, αν οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί, θα δημιουργηθούν ζημίες, ε, οπότε η συλλογική, η ομαδική θέρμανση θα πάψει να λειτουργεί, οι πολίτες θα επιστρέψουν στην ατομική θέρμανση και αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη μόλυνση. Οπότε θα πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Οι κανόνες, τα πρότυπα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά. υπέβαλα τροπολογίες που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι η οδηγία θα εξυπηρετεί και το περιβάλλον και τους πολίτες. Ευχαριστώ. Yes, thank you, Chair, and uh, thanks a lot. Ο κ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Θα είμαι σύντομος. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι τόσο κακή όσο θεωρεί ο εισηγητής. Βλέπω βέβαια κάποια πρακτικά προβλήματα τα οποία το Συμβούλιο τα επιλύει. Ιδιαίτερα τις εξαιρέσεις. Για παράδειγμα οι εξέδρες, οι θαλάσσιες εξέδρες και οι ε, επικαλύψεις με την ε, ε, οδηγία περί βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Είναι σωστό να χωριστούν αυτά τα δύο, αλλά όχι τελείως. Μόνο η ισχύς που ξεπερνάει τις, ε, τα όρια της MCP ε, θα πρέπει να εξαιρεθούν. Και αυτό είναι δύο μόνο περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλό που η συγγητής δέχεται πολλές προτάσεις του Συμβουλίου. Για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους. Δεν βλέπω όμως γιατί ο εισηγητής κάνει τόσο σημαντικές και τόσο πολλές αλλαγές στα παραρτήματα χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολύ λεπτομέρειες μελέτες για να καταλήξει αυτά τα νούμερα. Η αύξηση, η αλλαγή αυτών των αριθμητικών στοιχείων χωρίς ε, στοιχειοθέτηση δεν είναι σωστή. Βέβαια, αν έχουμε επιχειρήματα να, να τα συζητήσουμε, αλλά η γενική και σε βάθος αλλαγή των παραρτημάτων πιστεύω ότι είναι υπερβολική. Σε ορισμένες χώρες, όπως στις κάτω χώρες, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτή που προτείνει η οδηγία της μεσαίες, ε, μεσαίου μεγέθους. Για παράδειγμα, ε, μην ξεχνάμε, το 80% των καταστάσεων αυτών είναι καυστήρες. Από το 98% στις κάτω χώρες έχουμε εθνική νομοθεσία που διέπει ε, τους καυστήρες που βρισκόνται ε, που έχουν ισχύ χαμηλότερη από αυτή που προτείνει η οδηγία για τις μεσαίες μονάδες καύσης. Τώρα, ε, κάποιες από τις εξαιρέσεις για τις οποίες μίλησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, το Συμβούλιο προτείνει εξαίρεση για χίλιες ε, ώρες λειτουργίας. Όμως για μένα αυτό ανοίγει τη δυνατότητα οι εγκαταστάσεις αυτές να χρησιμοποιούνται χωρίς κανένα περιορισμό, δηλαδή όπως χρησιμοποιούνται τώρα. Να μην κρατήσουμε τις 500 ώρες και για τις βόρειες χώρες όπως Φιλανδία και σκανδιναβικές χώρες γενικότερα. Τι πιστεύετε η Κομισιόν για αυτό το θέμα. Μετά, ε, το πεδίο εφαρμογή και η ε, καταξινόμηση μια ακόμα ομάδα για, ε, τι, για τα 5-15 ΜΒ. Το κόστος είναι ψηλό από το 1 στα 5 ΜΒ και μετά το μειώνεται, αυτό το έχει πει το Συμβούλιο, μετά τα 5 ΜΒ το κόστος μειώνεται, οπότε δεν καταλαβαίνει να χρειαστούμε μία ακόμα κατηγορία μεταξύ 5 και 15. Γενικά, πιστεύω ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν είναι αρκετά ισορροπημένη και δημιουργεί ε, κανόνες υγιούς ανταγωνισμού. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας στόχη. Για να σας δείξω τι είναι δυνατό να γίνει ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να έρθει στην, ε, στις κάτω χώρες και να επισκεφθεί ε, μια ε, πολύ γνωστή ζηθοποιία των κάτω χωρών που ανακαίνισε τους καυτήρες ε, της δεκαετίας του 60 του 70 με σύγχρονη τεχνολογία και αυτή τη στιγμή έχει μειώσει τις εκπομπές σε κάτω από 70 μιλιγκράμμ διοξιδίου του αζότου. Ελάτε μια μέρα στις κάτω χώρες να δείτε αυτές τις εγκαταστάσεις. Κυρία Ροντρίγες Ρούβιο. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε για το θέμα της υγείας των πολιτών που πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Η κακή ποιότητα του αέρα κάθε χρόνο ε, προκαλεί 400.000 πρόορους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαιτέρως μάλιστα στην δική μου περιοχή, την Ανταλουσία, πάνω από το 90% του πληθυσμού ε, αναπνέει αέρα μολυσμένο παραπάνω από τα πρότυπα και τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πολύ δε περισσότερο που δημιουργούνται και προβλήματα στο οικοσύστημα. Ε, το κράτος δεν παίρνει μάλιστα μέτρα για να λύσει το πρόβλημα, οπότε πρέπει να το κάνουμε εμείς. Στο, ε, στα, τα προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση μόλι του αέρα πολλές φορές δεν υπάρχουν παρόλο που είναι υποχρεωτικά. Ή ακόμα και όταν υπάρχουν δεν εφαρμόζονται. Επιπλέον δεν ενημερώνεται αρκετά ο πολίτης. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λοιπόν την υποχρέωση να μεριμνήσουν έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Ε, η έκθεση αυτή όμως μερικές φορές κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει η αιτιολογική έκθεση. Να βρει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του πολίτη και να ε, περιορίσει το, το κόστος της επιχείρησης και τους ιδιώτες. Ε, αυτή τη στιγμή οι εξαιρέσεις είναι, δεν είναι αρκετά, ε, μάλλον αντιστοιχούν σε απόψεις που δεν είναι πολύ φιλόδοξες σε ό,τι αφορά την προστασία του πολίτη. Ε, ε δεν είναι δυνατόν να εξαιρούμε ε, τις εξέδρες εξόριξης στη θάλασσα, τις εγκαταστάσεις των νησιών ή χαρτοβιομηχανίες ως μεσαίες εγκαταστάσεις. Θα, με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε, χαμηλώνουμε τον πύχη αντί να τον αυξήσουμε. Η οδηγία δημόσιας υγείας ε, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο αυστηρή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ποιες είναι οι διαφορετικές ε, ε, τα διαφορετικά προβλήματα και αυτοί που ρηπαίνουν θα πρέπει να πληρώνουν. Οι οριακές τιμές εκπομπών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χαμηλές. Είναι χαμηλότερες ακόμα και από αυτές ορισμένων κρατών μελών όπως μόλις είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Για παράδειγμα, η Ολλανδική νομοθεσία είναι σαφής. Ε, έχει χαμηλότερα όρια εκπομπών, κάτι που οδηγεί σε βελτίωση της, ε, των καυστήρων. Με την τεχνολογία θα μπορούσαμε να μειώσουμε το 75%, ε, κατά 75% τις εκπομπές των οξυδίων του αζότου. Νομίζω ότι με χαμηλότερα όρια θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Από την άλλη μεριά η οδηγία προτείνει τη χρήση των ε, ε, εγκαταστάσεων ε, μέχρι το 2025, 10 χρόνια ακόμα λοιπόν. Η εφαρμογή των οριακών τιμών προτείνει οδηγία έρχεται καθυστερημένα ήδη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια. το προσχέδιο από την άλλη μεριά θεωρεί πως το αποτυχημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, αλλά με τη μείωση ε, των τιμών ε, δεν υπάρχουν πλέον κίνητρα για να μεταβούμε σε καθαρές μορφές ενέργειας. Επίσης, οι ιδεολογικές σκέψεις 2 και 3 δεν θεωρούμε ότι είναι σωστές. Ε, συγγνώμη, 12 και 13 δεν θεωρούμε ότι είναι σωστές και θα, υποβάλουμε πρόταση τροπολογίας. η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να δώσει το μήνυμα ότι ε, ε, παρακολουθούμε τις, την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Εμείς στην Ανταλουσία έχουμε σημαντικό πρόβλημα και παρακολουθούμε πολύ στενά το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you very much. And now, Madame Rivasi, can I ask to be short? Στο κυρία Ριβαζή, παρακαλώ να είστε λίγο πιο σύντομη γιατί 11 η ώρα θα έρθει ο Επίτροπος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Όπως ε, έχω ήδη πει, εμείς ε, οι οικολόγοι η ομάδα των οικολόγων υποστηρίζουμε πραγματικά αυτή την οδηγία όπως προτείνεται από την Κομισιόν. Και μάλιστα θα θέλαμε περισσότερο να προχωρήσουμε ακόμα σε σχέση με την ε, προστασία της ποιότητας του αέρα. Πρόκειται για τις μεσαίες οδηγίες, αλλά πρόκειται και για μια... Ε, με αλλά πρόκειται για θέμα η δημόσιας υγείας. Θυμηθείτε, 400.000 νεκροί ετησίως στην Ευρώπη. Πέρα από κάθε προβληματική δηλαδή που αφορά το κάπνισμα ή τα οδικά ατυχήματα τα αυτοκινητιστικά. Να πω κάτι όμως και να πάω κατευθείαν στο στόχο. Κύριε Σιγητά, όταν βλέπω τις εξαιρέσεις, ε, αυτή η οδηγία κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα. Βλέπουμε την τροπολογία 11. Εξαιρούνται οι ε, αεριοστρόβιλοι ε, ή πλωτές εξέδρες εξόριξης μετά ε, μετατροπή υδροθείου σε θείο. Έπειτα, εξαιρείται η χημική βιομηχανία. Έπειτα, εγκαταστάσεις για την κατασκευή καταλυτών κτλ. Κάμινοι, υψικάμινοι, κλίβανοι κρεματορίων κτλ και κερασάκι στην τούρτα, μέση καύση στα ε, Κανάρια, στα ε, ε στις Αζόρες και στα γαλλικά περπόντια διαμερίσματα. Μα δεν καταλαβαίνω. Αν αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου, ε, τα κράτη θέλουν να υποστηρίξουν ε, τα ο καθένα στο νομό του. Και εγώ είμαι Γαλλίδα και λέω ναι, ναι, πρέπει να προστατευτούν, μα ακριβώ εκεί πρέπει να υπάρχουν οι, καύσι, οι μονάδε που ε, σέβονται τι αρχέ. Εγώ είμαι κατά κάθε ε, εξαίρεση τέτοιου τύπου. Εάν επιθυμούμε να καινοτομήσουμε, να, να, να πιέσουμε του βιομηχάνου μα και ειδικά του Ευρωπαίου βιομηχάνου, ώστε να φτιάξουν μηχανέ που, να ε, που να ρηπαίνουν λιγότερο, πρέπει να το κάνουμε παντού. Ενώ άμα βρεθούν τα παραθυράκια, εκεί θα πάνε να στριμωχτούν όλοι. Ε, όχι λοιπόν, δεν ακολουθούμε το Συμβούλιο. Έπειτα, ε, οριακές τιμές. Είδα, έχετε τροποποιήσει τις οριακές τιμές τόσο όσον αφορά το διοξίδιο του θείου όσο και το μονοξίδιο του αζότου. Είμαι υπέρ των προτάσεων της Κομισιόν γιατί αν αυξηθούν οι οριακέ τιμέ, να είναι λιγότερο δεσμευτικέ, α πούμε. Γιατί να εισηχθεί έπειτα το 15. Η Κομισιόν είχε προτείνει 1 μέχρι 5 και 5 μέχρι 50 για ισχύ. Τι, γιατί να βάλετε ακόμα και το 15 στη μέση. Άμα θέλουμε να μειώσουμε κυρίως από το 5 έως το 50 είμαστε ήδη σε μεγάλες μονάδες. Και έπειτα υπάρχει μια τροπολογία για την οποία δεν έγινε πολλής λόγος. Αυτό το πρόβλημα της απόδοσης και της ε, ε, ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα κύριε ε, Σιγητά. Έχουμε τώρα ε, μονάδες κάθε βιομάζας που φτιάχνουν, παράγουν ηλεκτρικό. Ε, όμως πρόκειται για καύση ε, τεράστιων όγκων ξυλίας που δεν παράγουν καν ε, θέρμανση. Υπάρχουν όλα ένα περισσότερες στις ευρωπαϊκές, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Δηλαδή εντάξει να φτιάχνουν ηλεκτρισμό με το ξύλο, αλλά τουλάχιστον να ανακτούν τη θερμότητα πέρα από το 60-70% γιατί διαφορετικά πάνε τα δάση για να φτιαχτεί μόνο ηλεκτρισμός ενώ η, ζέστη φεύγει στην ατμόσφαιρα. Μα είναι φρικτό αυτό. Υπάρχουν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν λοιπόν στο κείμενο. Ε, πρέπει μια θέση των ε, οικολόγων είναι να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε λιγότερες εξαιρέσεις γιατί διαφορετικά όπως είπα θα μείνει καινογράμμα και έπειτα να προχωρήσουμε στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ τελευταίος ομιλητή της Πελιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία που έκανε μέχρι στιγμής, για το σχέδιο έκθεσης. Ε, και αν σκεφτούμε την αβεβαιότητα για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Juncker για το 2015 σε σχέση με το καθαρή ατμόσφαιρα. Εμείς συμφωνούμε με όλα, μόλις, με όλα όσα μόλις είπε η συνάδελφος Ριβαζή και η Πράσινη όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τις οριακές τιμές στο κείμενο. Έπειτα η πρόταση της οδηγίας δεν θα πρέπει μόνο να ε, συνδυάζεται με την 2009 ε, για το σχεδιασμό και αυτή του 2010 για τις εκπομπές ε, ρήπων. Θα πρέπει να επιμείνει και για τη τεχνολογία που είναι φιλική προς το περιβάλλον, να προβλέψει την πρόσβαση στις αγορές των πιο καλών ε, τεχνολογιών που βρίσκονται στην αγορά, να σεβαστεί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που επιτρέπουν μόνιμες προδιαγραφές αποτελεσματικές όσον αφορά το κόστος, αλλά και όσον αφορά τον καθαρό αέρα Λογικό επίσης, λογική επίσης ε, εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και προστασία της ποιότητας του αέρα. Ο έλεγχος και διαρκής που θα, θα είναι εγγυημένος από τρισδιάστατους καταμετρητές που διαβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο ε, τα στοιχεία στην αρχή διαχείρισης. Έτσι ε, όπως ζητήθηκε και από την Επιτροπή Αόρος, αλλά και από την, το, το, άρθρο περί των βιομηχανικών εκπομπών, της οδηγίας μάλλον περί βιομηχανικών εκπομπών. Θα πρέπει να εγγυηθούμε λοιπόν καθαρό αέρα και ασφαλή παντού, ξεκινώντας από τις μικρές και μεσές ε, μονάδες. Δεν θα πρέπει ωστόσο να μείνει ατελής, γιατί ε, εκεί ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρόκειται την, για τη γενιά μικροτρή που επιτρέπει την διάχυτη διάδοση. Ευχαριστώ να δώσω σύντομα το λόγο στον κύριο Τάνς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το μισό πακέτο ποιότητα στο αέρα, το άλλο μισό βεβαίω είναι οι εθνικέ οροφές ε, και μια που είμαι εισηγητή, εγώ στο άλλο μισό νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι κάνουμε και εδώ πέρα. Και πρέπει να πω πω απογοητεύτηκα λίγο, εγώ συμφωνώ πλήρω με τον κύριο Παλούτσι όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξία. Ε, της έκθεσης αυτής. Γνωρίζουμε την κλίμακα του προβλήματος, ε, το συζητάμε συνέχεια, αλλά δεν έχει νόημα να πάμε με μια διαπραγματευτική θέση απέναντι στο Συμβούλιο και να έχουμε την ίδια θέση ή ακόμη και πιο εξασθενημένη. Πρέπει να είμαστε σαφείς ε, ως Κοινοβούλιο τι θέλουμε, τι επίπεδο φιλοδοξίας έχουμε και με αυτή την βάση νομίζω πως όπως ήδη υπόθηκε το, τα επίπεδα των εξαιρέσεων και όλα τα υπόλοιπα νομίζω εξασθένησαν μια σημαντική έκθεση. Η τεχνολογία υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος λοιπόν για αυτές τις εξαιρέσεις για τα μεσαίου, για τις μεσαίου μεγέθους ε, μονάδες ε, και απευθύνω έκκληση και για αυτό το νομοθέτημα να είναι εξίσου νομοθέτημα γιατί τελικά θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα εάν ε, λειτουργήσουμε οργανωμένα στο επίπεδο που προτείνει η Κομισιόν. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το ελάχιστο σαφετήρια. Ευχαριστώ. Κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχα αρκετά πράγματα, θα περιοριστώ σε έναν. Αναρωτιέμαι γιατί αντικαταστάθηκε η λέξη σωματίδια με τη λέξη σκόνη στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω. Η σκόνη δεν είναι επιστημονικός όρος, ενώ τα μικροσωματίδια καλύπτει πλήρως αυτό το οποίο εννοούμε. Χρησιμοποιείται σε όλη την νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εισηγητή γιατί άλλαξε αυτή τη λέξη και έγραψε σκόνη. Ευχαριστώ. Κύριος Λίντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις εγκαταστάσεις μεταξύ ενός και 5 ΜΒ και ειδικά αυτές που καίνε βιομάζα και ξύλα ειδικά στην πατρίδα μου έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να λεφθούν υπόψη γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν και να ανακαινιστούν αυτοί οι καυστήρες και αυτοί οι καταστάσεις εκ των υστέρων. Όταν αγοράζει κανείς λοιπόν μια συσκευή που κοστίζει 200.000 ευρώ είναι μια μεγάλη επένδυση και νομίζω είναι σαφές μετά πως είναι δύσκολο να την ε, ξαναλλάξει αν δεν έχει γίνει μία απόσβεση και τελικά τι θα κάνει θα αντικαταστήσει το καύσιμο με ορυκτά ε, καύσιμα αυτά σας ευχαριστώ δίνω τώρα τον λόγο για ένα σύντομο σχόλιο στην Κομισιόν στον κύριο... Α, με συγχωρείτε, ο κύριος Χέλνερ. Ναι, ναι, θα είμαι Είναι σημαντικό αυτό το νομοθέτημα για να φτάσουμε στους εθνικούς στόχους. Το μόνο το οποίο μας ε, ανησυχεί είναι οι μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν ε, στέρεα βιομάζα, ειδικά αν μιλάμε ας πούμε για ε, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξυλίας δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η δασοκομεία ε, ειδικά για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οπότε πρέπει νομίζω να μην, ε, πρέπει να μην ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία θα κλείσει τις μικρές τέτοιες ε, επιχειρήσεις. Γιατί τελικά θα οδηγηθούμε σε περισσότερες εισαγωγές, σε περισσότερες μεταφορές που θα βλάψουν το περιβάλλον. Ε, ανησύχησα κάποια πράγματα όπως ε, η επικάλυψη, τα είπε αυτά ήδη ο εισηγητής, ε, οι ώρες λειτουργίας επίσης δεν θα πρέπει να καθιστούν αδύνατη την λειτουργία τους. Το μόνο στο μέσο με είναι ακριβώς τα για τις μικρές εγκαταστάσεις βιομάζας, ειδικά για τα σωματίδια. Δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε τώρα το όριο ή την ε, οδηγία αυτή για τις βιομηχανικές ε, εκπομπές, όπου έχουμε κάποιες εξαιρέσεις για την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, αν παραδείγματος χάρη η γεωγραφική θέση σημαίνει πως δεν ε, υπάρχουν άμεσες συνέπειες από τα σωματίδια για ανθρώπους ή για το περιβάλλον. Ή αν για τεχνικούς λόγους δεν γίνεται κάτι. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση λοιπόν όπου δεν έχουμε επίπτωση στο περιβάλλον αλλά έχουμε τεράστιο κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο χαλεμ ε, Σας παρακαλώ να είστε σύντομος γιατί Περιμένει ο Επίτροπος να ε, έξω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα και σημειώνουμε με ικανοποίηση πως υποστηρίζεται ε, εδώ πέρα η θέση του εισηγητή πως το πεδίο εφαρμογή ε, από το 1 στα 50 ΜΒ πρέπει να διατηρηθεί και πρέπει να ασχοληθεί και με τη γενική ρήπανση, αλλά να δίνει και μια κατεύθυνση στα κράτη-μέλη για το πώς ασχοληθούν με κάποια πάρα πολύ έντονα σημεία. Εδώ πέρα όμως ανησυχούμε πως ε, το να κατεβάσουμε το παράρτημα 3 στα επίπεδα των νέων ε, μονάδων δεν ε, ανταποκρίνεται στις πιο προχωρημένες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ισχύσουν σε τέτοια επικίνδυνα σημεία ρήπανσης. Αυτό το οποίο είχαμε προτείνει εμείς νομίζουμε πως ήταν μια καλή ένδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί και αν το εξασθενήσουμε θα στείλουμε λάθασμένο μήνυμα στην βιομηχανία ένα κλάδο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ηγετικό ρόλο και θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις ΙΠΑ ή τους ανταγωνιστές στην ΑΠΟ Ανατολή αν δεν παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή. Ανησυχούμε για το ότι κάποιες διατάξεις λοιπόν έχουν εξασθενήσει γιατί η πρόταση που έχουμε υποβάλει εδώ πέρα έχει σχεδιαστεί να είναι κάτι το οποίο θα μπορούν να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προσφέρει μια μακροπρόθεσμη σιγουριά με το 2025 ως προθεσμία και εάν είναι πάρα πολύ εξασθενημένα εξασθενημένες οι διατάξεις θα χρειαστεί να τις αναθεωρήσουμε σε λίγα χρόνια και έτσι θα πάνε χαμένες ε, οι επενδύσεις. Η καθυστέρηση επίσης κάποιων διατάξεων είναι προβληματική προβλέπουμε πάλι και μία μακροπρόθεσμη πολιτική μέχρι το 2030 και κάποιες εξαιρέσεις μέχρι το 2035. Έτσι δεν θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη λοιπόν να ε, επιτύχουν ε, ένα αποδεκτό επίπεδο καθαρό αέρα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Και επίσης σημειώνουμε γιατί υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις για το παράδειγμα 2 να αναφέρουμε τις ε, ανησυχίες που τονίσαμε και στο Συμβούλιο. Βλέπουμε πως ε, υπάρχει εδώ πέρα μια υποχώρηση ειδικά στο θέμα του θείου. Υπάρχουν κάποια καύσιμα με υψηλό περιεχόμενο θείου, θέλουμε να χρησιμοποιούνται, γι' αυτό χρειάζεται, χρειάζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Κάποιες από τις τροπολογίες λοιπόν που προτείνονται Ε, ε, μεταθέτουν το στόχο στο 2025 στόχο μείωσης του θείου και έτσι θα επηρεαστούμε πάρα πολύ από τα σωματίδια που ανασένουμε στις πόλεις μας. Όσον αφορά την ε, παράλληλη νομοθεσία, πράγματι συμφωνούμε και υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη χάρτοβιομηχανία και τα διελιστήρια θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια συμμόρφωση με την οδηγία για επαγγελματικές, για βιομηχανικές, με συγχωρείτε αλλά προσέξτε, στην τροπολογία μην καταλήξουμε οι μεγάλες βιομηχανίες να έχουν πιο ευνοϊκό καθεστώς ε, από τις ε, μικρομεσές. Αυτή είναι η μόνη μας επιφύλαξη. Αυτά ήταν τα σχόλια που είχα να κάνω κύριε Πρόεδρε, να αναφέρθηκα σε, κάποια, σε κάποιες ερωτήσεις που απευθύνθηκαν συγκεκριμένα προς την Κομισιόν. Αν θέλετε μπορώ να επανέλθω ή δίμερος. Τέλος, ζητώ συγγνώμη, ο διευθυντής μου ή διευθύντρια ήθελε να έρθει σήμερα, αλλά αρρώστησε, δεν είχε την δυνατότητα. Τελευταίο, τελευταίο σχόλιο, ο κύριος Γκρίβης, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Τα μέλη, αγαπητοί σκιοσυγητές. Δεν ήταν επιδενή πρόθεσή μου να αποδυναμώσω την νομοθετική πρόταση. Αξίζει όμως να υπογραμμίσουμε ότι κάθε μία από τις προτάσεις μου έχει μία αιτιολόγηση. Βασίζεται σε έγγραφα τα οποία ε, διαθέτουμε και είναι ανοιχτό να σας εξηγήσω και να καταλάβω και ενδεχομένω και τις δικές σας αντιρρήσεις όταν έχετε. Στην περιπτώση, σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, με, πολλές, με πολλά διαμερίσματα, με κεντρική μονάδα καύσης για τη θέρμανση, θα πρέπει να αποφύγουμε να θέσουμε σε αυτές τις μικρές εγκαταστάσεις, να θέσουμε στις μικρές εγκαταστάσεις ε, πιο αυστηρούς όρους. Γιατί αν θέσουμε αυστηρούς όρους για αυτούς τους κεντρικούς καυστήρες, ε, οι καταναλωτές θα απομακρυνθούν από τη χρήση τους και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν ατομικούς καυστήρες. Αυτό το έχουν δει Δεν είναι κάτι καινούριο που λέω. Γι' αυτό το λόγο θέλω να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Όπως είπα, Είμαι πρόθυμο να τα συζητήσω όλα αυτά. Έχουμε όμω χρονικό περιορισμό, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν μπορώ να σχολιάσω καθένα, κάθε μία από τι παρατηρήσει σα. Η Κομισιόν είναι εδώ. Ε, δεν θα κάνω ποτέ άλλο παρά να ευχαριστήσω ε, όλου του συναδέλφου για την ανταποκριτική του σχόλια. Πρόεδρο. Οι προθεσμοί για τι τροπολογίε με ψηφιακή υπογραφή λίγη στι 5 Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι. Ε, η τροπολογίες θα συζητηθούν στι τελευταίε συνεδρίε του Μαρτίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 13 ή 14 Απριλίου. Το σημείο 7 τη ε, ημερήσεω διαταξή μα θα συζητηθεί μετά τι ψηφοφορίε της ε, απογευματινής μας συνεδρίασης. Οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν ε, στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Καρμένου Βέλα, Επίτροπο Ερμόνιο του Περιβάλλον, Θαλάσσια Πολιτική και την Αλία. Χαρά μου είναι να σας, που σας έχουμε εδώ μαζί σήμερα, κύριε Επίτροπε. Ας ξεκινήσουμε αμέσω τη συζήτηση. Ε, το όπως γνωρίζετε έχουμε πολλές προσδοκίες από εσάς και από τη, για τις δραστηριότητε σας ε, τα, επόμενου μήνε. μήνες. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα σας θέσουμε ερωτήσεις. Αργότερα βέβαια θα απαντήσετε και εσείς όπως πάντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Τζοβάνι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλα τα μέλη. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας ε, που με καλωσορίζετε σήμερα στο Κοινοβούλιο για μια ανταλλαγή απόψεων για τις ε, προτεραιότητες μας για φέτος αλλά και γενικότερα για τους ε, στόχους κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου είχα υποσχεθεί να είμαι ανοιχτός και να διαφανίσαι μπροστά σας. Από όταν ξεκίνησα την 1η Νοεμβρίου ήδη συνάντησα πολλούς από εσάς και πολλές από εσάς διμερώς. Η γνώμη σας ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για μένα. Και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι ένα ακόμα βήμα για την ανάπτυξη αυτού του διαλόγου μεταξύ μας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μου είχα λάβει δέσμευση να είμαι προσιλωμένο στο 7ο πρόγραμμα, περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης. Το δικός χάρτης αυτού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κινηθούμε προς μια οικονομία πιο καινοτόμα, χαμηλές ε, άνθρακα ε, και ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε το φυσικό μας κεφάλαιο, την υγεία και την ευμερία των πολιτών. Σήμερα θέλω να σας υπογραμμίσω το πώς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον οδικό χάρτη ως Κομισιόν για το 2015. Ας ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν και το οποίο έχω ήδη συζητήσει με αρκετούς από εσά τις περασμένες εβδομάδες. Είναι η κυκλική οικονομία, το πακέτο για την κυκλική οικονομία συγκεκριμένα. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εσά εδώ στην Επιτροπή διαφωνούν με την απόσυρση της αναθεώρησης νομοθεσίας περί αποβλήτων. Ε, ξέρω επίση ότι είσαστε διστακτικοί σε ό,τι αφορά τι υποσχέσει μα να υποβάλουμε μια πιο φιλόδοξη πρόταση φέτο. Κατανοώ ότι ίσω υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί, αλλά θυμηθείτε παρακαλώ ότι έχουμε αναλάβει τη δέσμευση και αυτή η δέσμευση θα υλοποιηθεί. Η Κομισιόν θα ολοκληρώσει την απόσυρση ε, τις επόμενες μέρες. Τώρα θα εστιαστούμε λοιπόν στην υποβολή νέων προτάσεων που θα πρέπει να έχουν γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, στην καινούρια πρόταση. Το κίνητρο μας είναι απλό. Θέλουμε να βάλουμε την Ευρώπη σε ένα μονοπάτι προς ένα πραγματικό γνήσιο, ε, προς μια πραγματικά γνήσια ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την κυκλική οικονομία αλλά και να ε, ε, αποσύρουμε όποιες αβεβαιότητες υπάρχουν στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά ε, τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασία που πρέπει να δημιουργηθούν. Το κείμενο στο πρόγραμμα εργασία μας είναι σαφέστατο. Απόσυρση και αντικατάσταση με νέα πρόταση μέχρι το τέλος του 2015 για να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία. Δεν υπάρχει εκεί καμία αμφισημία. Οπότε, το κίνητρο μας είναι σαφές, ο στόχος μας είναι απλός. Ε, όμως, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Αυτή η προσέγγιση είναι δυτή. Πρώτον, θέλουμε να υποβάλουμε μια καινούργια νομοθετική πρόταση σε ό,τι αφορά τους στόχους για τα απόβλητα. Αυτή η νέα πρόταση θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που έχουμε ήδη συλλέξει κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα τα σχόλια που έγιναν από Πολλού που έλεγαν ότι οι προτάσει για τα απόβλητα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένε. Η Κομισιόν θα εξετάσει όλε τις καινούριε πληροφορίες, αλλά θα βασιστεί και σε παλιότερε εργασίε που είχαν γίνει για την προετοιμασία τη προτάσεω για τα απόβλητα. Θα ήθελα να σα. καθισκάσω. Η νέα πρόταση θα διατηρήσει το όραμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων και για τον στόχο τη αύξηση ε, των ποσοστών ανακύκλωση στην Ευρώπη. Χρειάζεται να θέσουμε αποτελεσματικούς, ε, εφιλόδοξους και ε, ευφύς Η επιτυχία μας θα μετρηθεί από το πόσο καλά θα εφαρμόζονται οι πολιτικές μας σε κάθε κράτος μέρος. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Δεύτερον, θα κλείσουμε τον κύκλο της κυκλικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι θα εξετάσουμε την βιώσιμη κατανάλωση αλλά και παραγωγή. Και ανάντι την παραγωγή και την φάση χρησιμοποίηση, δηλαδή πριν τα προϊόντα γίνουν απόλυτα, αλλά και κατάντι, δηλαδή αφότου τα προϊόντα πάβουν να είναι απόλυτα πλέον. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε και να αναπτύξουμε μια αγορά για τα ανακυκλωμένα προϊόντα. Αυτό που η έκφραση που έρχεται στο μυαλό μου είναι χρησιμοποίησέ το ή θα το χάσεις. Θα ήταν πραγματικά ηρωνικό να ε, καταναλώσουμε σημαντικές προσπάθειες ε, για να δημιουργήσουμε ανακυκλώσιμο, ε, επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και τελικά να μην τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό έτσι κοιτάμε εμείς το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα ανακυκλωμένα υλικά θα ξαναμπούν στην παραγωγική αλυσίδα. Με παρόμοιο τρόπο η ανακύκλωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί, να γίνει πιο οικονομική και πιο αποτελεσματική αν τα προϊόντα σχεδιαστούν ήδη εξ αρχής και χρησιμοποιηθούν με το στόχο της μείωσης των αποβλήτων. Ο, αυτό είναι το άλλο μισό του κύκλου, έτσι το ονομάζουμε εμείς και θα το δείτε με σάρκα και οστά στον οδικό χάρτη όπου θα εντοπίζουμε ακριβώς ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Επίσης, εξετάζουμε can to our... το πώς ε, η κυκλική οικονομία μπορεί να συνεισφέρει στους στόχους μα περί ενεργειακή αποδοτικότητας. Ε, μια πτυχή στην οποία θα αναφερθεί και ο, πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς ε, ε, στο, στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή την Ενεργειακή Ένωση που θα παρουσιάσει αύριο στην Ολομέλεια. Και οι δύο πλευρές αυτού του πακέτου θα είναι έτοιμες μέχρι το, 2000, μέχρι το τέλος του 2015. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε πως ε, πρόκειται για ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραμμα σύμφωνα με το 7ο ε, πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον και ε, σύμφωνα επίσης με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη στους οποίους θα επανέλθω σε λίγο. Να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος 12 των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΕΕ αναφέρει διτά ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το πακέτο αποβλήτων από μόνο του δεν θα μας έδινε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Ας εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό την πρόκληση από κοινού, μαζί. Το να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αξία των πόρων που διαθέτουμε απαιτεί δράση σε όλα όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Από την εξαγωγή των ε, πρώτων υλών στην, ε, ε, στο σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των αγαθών, στην επισκευή, στην επαναχρησιμοποίησή τους, στην διαχείριση των αποβλήτων και πάλι την ε, επιστροφή στην αλυσίδα παραγωγής. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, έχουμε συλλέξει απόψεις για την πρόταση περί αποβλήτων που παρουσιάσαμε το περασμένο καλοκαίρι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά ειλικρινά όλους και όλες εσάς για το ενδιαφέρον που δείξατε και πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε και στο μέλλον. Επίσης, ε, θα καθορίσουμε, έχουμε ήδη μια σειρά δράσεων, εργαλείων και μέτρων ε, στις τομείς ε, που αφορούν τα προϊόντα και τα, τις χημικές ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν στην κυκλική οικονομία. Θα πρέπει να συγκεράσουμε όλη αυτή την γνώση μαζί με την πολιτική μας βούληση για έτσι ώστε το πακέτο να είναι όσο πιο φιλόδοξο γίνεται. Το περασμένο Δεκέμβρη στη Λιόν είδα εξαιρετικέ ε, εξαιρετικές ικανότητες ε, οικολογικής καινοτομίας στην, ε, στην απονομή των βραβείων ε, ε, περιβάλλον, περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη δημιουργικότητα ακόμα περισσότερο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, εργαλεία όπως η οδηγία για την, την οικολογικό σχεδιασμό έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, κυκλική οικονομία ε, και τι θα κάνουμε με την ποιότητα των ανακυκλωμένων προϊόντων. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία περιχημικών για να βελτιώσουμε την ποιότητα και να αποφύγουμε χημικές ουσίες που είναι βλαβερές να επιστρέψουν στην αλυσίδα της παραγωγής. Και τι θα γίνει με, τα κρίσιμα, με τις κρίσιμες πρώτες ύλες η βιομηχανικά, τα βιομηχανικά απόβλητα αντιστοιχούν στο 50% των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι καλύτερε διαθέσιμες τεχνικές για να βελτιώσουμε την ε, βιομηχανία της κυκλική οικονομίας. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ε, και τι γίνεται με μια πολιτική καταναλωτή που θα εστιάζει περισσότερο στην, στους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την κυκλική οικονομία μέσω χρηματοδοτικής στήριξης. Αυτές όλες είναι ερωτήσεις που χρειάζεται όλοι μαζί να απαντήσουμε στους επόμενους μήνες. Τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να συνδυάσουν νομοθετική δράση, ε, μέτρα, μάλλον ε, εργαλεία που βασίζονται στην αγορά, έρευνα και ανάπτυξη, κίνητρα, ανταλλαγή πληροφοριών ε, και εθελοντικής φύσεως προσεγγίσεις. Όλα αυτά θα δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα στις επιχειρήσεις εργαλεία τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Η ε, Κομισιόν ετοιμάζει μια ε, εισαγωγική έκθεση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στρατηγικών Επενδύσεων και εκεί υπογραμμίζει ε, τη σημασία της ε, αποδοτικής χρήσης των πόρων που είναι ένας βασικός στόχος. Αυτό θα πρέπει να, αυτός ο στόχος θα πρέπει να γίνει ε, project ε, οικολογικής καινοτομίας ε, και να χρημα, θα χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά τα ταμεία. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα εργαλεία. Η δική σας άποψη θα είναι χρησιμότατη και όπως πάντα περιμένω να την ακούσω ήδη από σήμερα και μέσω της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για την κυκλική οικονομία που από ό,τι κατάλαβα μπορεί να, να εγκριθεί στην Ολομέλεια πριν το καλοκαίρι. Ας είμαστε λοιπόν πιο καινοτόμοι, πιο στρατηγικοί και πιο φιλόδοξοι όλοι μαζί. Σε ό,τι αφορά την προτινόμενη οδηγία για τις, για τις εθνικές οροφές εκπομπών είναι πολύ σαφές ότι παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα υποβάλουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μια τροποποιημένη πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις εξελισσόμενες θέσεις ε, των συνομοθετών ε, έτσι ώστε ε, να προωθήσουμε από κοινού την ενεργειακή πολιτική και την κλιματική πολιτική, να εστιάσουμε στην μείωση του γραφειοκρατικού βάρους χωρίς όμως να υποχωρούμε έναντι των αρχικών στόχων. Ε, τώρα έχουμε πλέον το εκτιμόμενο κόστος ε, που βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία, ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσαν τα κρατημέλη και μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Αναγνωρίζουμε ότι υφίστανται ακόμα ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, πτυχές της πρότασης και θα πρέπει να το δούμε. Αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών. Περιμένω την άποψη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση και σας ε, βεβαιώνω ότι εμείς ε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική και γρήγορη συμφωνία. Μόλις συζητήσατε την, ε, το προσχέδιο έκθεσης του κυρίου Γκζιμπ για τα, τις εγκαταστάσεις καύσης μεσαίου μεγέθους. Ζητώ συγγνώμη με το όνομά σας κύριο Γκριμπ, αλλά δεν μπορώ να το προφέρω πολύ καλά. Αυτές οι εγκαταστάσεις συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ε, μόλυνση του αέρα ιδιαίτερα σε αστικέ περιοχέ. Χαίρομαι που βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία πρώτη ανάγνωση με την Λετωνική Προεδρία. Η Κομισιόν θα διευκολύνει μια τέτοια συμφωνία. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για να πετύχουμε τους συνολικούς στόχους εκπομπών. Τώρα, περνάω ε, σε ένα άλλο θέμα μια άλλη πρωτοβουλία του προγράμματος εργασίας ε, με το οποίο ήδη έχουμε αποτελέσματα. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, με το, με το συνάδελφο Μίμικα ε, έχουμε υποβάλει, υποβάλαμε πριν από τρεις εβδομάδες μια ανακοίνωση για την εκκρίωση της ε, φτώχειας και την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Σεπτέμβρη φέτος οι κρατών κυβερνήσεων ζήτησαν ε, θα, μάλλον συγγνώμη, θα τους ζητηθεί να συμφωνήσουν στο πρόγραμμα πλαίσιο για μετά το 2015 ε, που θα ξεπερνάει και τους ε, στόχους χιλιετίας για την ανάπτυξη και θα υλοποιεί το, το αποτέλεσμα της διάσκεψης 2 20 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η, το ανακοίνωση αυτή θα καθορίσει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι απαραίτητο για να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ένα από αυτούς τους στόχους είναι η παραγωγή και κατανάλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ηγέτητα δύναμη σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον εντοπισμό νέων ε, κύκλων, βιώσιμων, κύκλων βιώσιμης ανάπτυξης και κατανάλωσης, ε, στην διακυβέρνηση των ωκεανών και στην προστασία των θαλάσσιων πόρων μας και των παγκόσμιων οικοσυστημάτων. Όπως γνωρίζετε από την ακρόασή μου, η διακυβέρνηση των ωκεανών είναι μία από τις ε, ε, προτεραιότητες της ε, θητείας μου. Η, ανακοίνωση που υιοθετήσαμε καθορίζει το όραμα της Κομισιόν για το τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί αυτή η ατζέντα. Περιέχει ιδέες για την παρακολούθηση, τη λογοδοσία και την αναθεώρηση των ε, μας μια σειρά από δράσεις θα καθορίσει το δρόμο προς την εφαρμογή του πλαισίου μετά το 2015 μέσω συγκεκριμένων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων. Αναμένω να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο αυτό το θέμα έτσι ώστε οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν ε, ε, επιτυχής δράση μέσω της ε, εφαρμογής ατζέντα για το, τη μετά το 2015 εποχή. Περνάω στην φυσική πρωτεύουσα ε, ε, ε, συγγνώμη, για το έτος φυσικής πρωτεύουσας, του φυσικού κεφαλαίου. Το 2015 είναι έτος προστασίας φυσικού κεφαλαίου και για να γίνει αυτό ε, να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε το, ε, το, καλό, την άνοιξη ε, με την νομοθεσία περί αποτελεσματικότητα, με την, τον έλεγχο της νομοθεσίας, και με την διάμεση έκθεση για την στρατηγική βιοποικιλότητας. όλα αυτά θα μπουν στο συνολικότερο πρόγραμμα αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέσω του πρόγραμματος REFIT. Ε, πολλοί από εσά, αλλά και πολλοί πολίτε και μη κυβερνητικέ οργανώσει δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην νομοθεσία περί φύση. Ε, η ε, Κομισιόν γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές, πολλά ευαίσθητα θέματα που σχετίζουν με το refit. Η Κομισιόν θα κάνει αυτή την αξιολόγηση με έναν τρόπο διαφανή και σφαιρικό θα είναι μια ευκαιρία να πάρουμε τις νόμες όλων ε, σε ε, εκδηλώσει όπως η Πράσινη Εβδομάδα στην αρχή του Ιουνίου που θέτως θα εστιάσει στην φύση και την βιοποικιλότητα καθώς επίσης και στην διάσκεψη των ενδιαφέρον μερών για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της νομοθεσίας το Σεπτέμβρη. Ε, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βασιστούμε και στη δική σας άποψη ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε την κοινή μας ατζέντα σε όλα αυτά τα θέματα ε, και ε, όταν θα συντάξουμε τα πορίσματα από τις έκθεσεις για το, την κατάσταση του περιβάλλοντος. Να πω όμως και δύο λόγια για το θέμα της εφαρμογής. στην ακρόση μου είπα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους και μάλιστα πολλές, σε πολλές περιπτώσεις να βελτιώσει σημαντικά τις αποδόσεις τους. Γνωρίζω ότι είναι κοινό μας ο στόχος για πλήρη ε, και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας που υιοθετείται σε συναπόφαση με το Κοινοβούλιο και γνωρίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν έχει νόημα να, έχουμε, να καθορίζουμε στόχους αν αυτοί δεν πληρούνται αργότερα δεν υλοποιούνται. Για να το πετύχουμε αυτό θα εργαστώ πιο στενά με τα κράτη-μέλη για να βοηθήσω να καταργήσουμε τους φραγμούς, να μάθουμε ποια είναι τα προβλήματά τους και να προωθήσουμε τη συμμόρφωση. Και εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό. Ε, θα σας ζητούσα να χρησιμοποιήσετε τα δίκτυά σας και την επιρροή σας, ο καθένας και καθεμία στη χώρα του έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην σωστή και πλήρη εφαρμογή. Αυτό θα οδηγήσει και σε πιο υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεών μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα διασφαλίσει ε, ψηλότερα ε, περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία αξίζουν οι μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αναμένω τα σχόλια και τι ερωτήσεις σα. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση και για το όραμά σας. Ζητήσαμε κάτι τέτοιο βεβαίως από την Κομισιόν και τώρα ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε τον Πίτερ Λίζε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα δώσω λόγο στον Λίγο Μπέλετ που είναι ο αρμόδιος ε, συντονιστής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Πέτερ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις βεβαίως. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το ότι η πρόταση ακόμα επιτάπτος και είπατε πως ακόμα θα καταθέσετε δύο προτάσεις. Θέλουμε βεβαίως μια πρόταση φιλόδοξη η οποία θα οδηγήσει σε ελάχιστη γραφειοκρατία. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε ε, το συγκεκριμένο αυτό παράδοξο όταν μιλάμε για τις εθνικές οροφές εκπομπών. Επιπλέον ξέρετε πως πάρα πολλά κρατημέλη ήδη έχουν δυσκολίες με την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων. Πώς θα βοηθήσετε τα κράτη-μέλη που δυσκολεύονται ήδη να επιτύχουν τους πιο φιλόδοξους στόχους στο μέλλον. Δεν είναι εύκολο. Τέλος, ε, να αναφερθώ στις προδιαγραφές κομπών ε, οχημάτων. Ξέρουμε πως ο κύκλος δοκιμών ε, που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στις εκπομπές του, τις πραγματικές. Υπάρχουν σχέδια να επανασχεδιαστεί αυτός ο κύκλος, αλλά τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε το 2017, τρία χρόνια μετά την υιοθέτηση των προδιαγραφών Euro 6 ε, να χρησιμοποιηθούν κάπως πιο ρεαλιστικοί κύκλοι δοκιμών. Ευχαριστώ Ματίας Κρότε για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ε, σε αντίθεση με τους ε, φίλους του ΕΛΚ εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι η Κομισιόν απέσυρε το πακέτο. Η ελπίδα βεβαίω πεθαίνει τελευταία. Ελπίζουμε να υπάρξει μια βελτίωση της κατάσταση Θα δούμε τι θα γίνει τι επόμενε μήνες και τι επόμενε εβδομάδες και μήνες. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος, να μην μείνουν τα πράγματα στην ε, μέση. Μην ξεχνάμε πω όσον αφορά τα απόλυτα και την ανακύκλωση και καθώς ε, και η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν είπε πως υπάρχουν ε, πάρα πολλές δυνατότητες και όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέχρι και 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Οπότε θα έλεγα πως δεν ναι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αναβολή αυτή. Αλλά εάν τελικά όντως καταλήξουμε σε μια καλύτερη πρόταση από την τωρινή τότε ευχαρίστως να την δεχτούμε. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, συχνά εμείς εδώ πέρα νομοθετούμε και νομοθετούμε συχνά αλλά βεβαίως η εφαρμογή πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη και εκεί ακριβώς είναι το ζήτημα γιατί συχνά τα κράτη δεν κάνουν αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε θα αναφέρω εγώ μόνο στην, στους βιότοπους Πανίδας και Χλωρίδας, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Αυτά τα οποία λοιπόν συμβαίνουν συχνά είναι πως ε, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, αποφασίσαμε από τον Ιανουάριο να εστιάσουμε στην εφαρμογή και βεβαίω αυτό σημαίνει ελέγχους και λεφτά για ελέγχους. Είστε αρμόδιος ε, και για την αλληλεία και εδώ πέρα όλα τα κράτη-μέλη κάνουν λίγο τα στραβά μάτια. Δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Χρειάζεται μια άλλη στρατηγική. Εδώ πέρα το 7ο πρόγραμμα δράσης έχει πει πως οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι έχει να μας πει η Επιτροπή για αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας και αν ε, εφαρμοστούν ε, στην πράξη νομίζω θα έχουμε καλά αποτελέσματα αλλά όπως είπα θα περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ για τους Ευρωπαίους Συντελετικούς κυρία Κέρλινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τις προσπάθειές σας ε, σιωπηρές συχνά για να παραμείνει ε, στο προσκήνιο το θέμα της ποιότητας του αέρα. Εγώ θα ήθελα να φέρθω τώρα σε κάτι άλλο για την οδηγία για τα πτηνά και τους βιοτόπους. Δεν την αναφέρατε. Έχουμε δει μια αρχική σας επιστολή, επιστολή του Πρόεδρου Γιούνκερ, στην οποία ζητάει να Αξιολογήστε ξανά το πώς ε, λειτουργεί αυτή η οδηγία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι γίνεται κάτι τέτοιο, προφανώς δεν μπορείτε να μας δώσετε μία οριστική απάντηση, αλλά θα ήθελα να μάθω πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και να μας διαβεβαιώσετε πως οι προτάσεις, οι τελικές δεν θα είναι αυτό το οποίο υποθέτουν πολλοί ότι δηλαδή θα έχουμε μια εξασθένηση της ε, προστασίας. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους ο κύριος Γκερμπράντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε. Πριν και κατά την διάρκεια της ακρόασης σας είχα προειδοποιήσει πως ε, θα ξεκινήσατε με μάχες, κάτι το οποίο αποδείχθηκε ε, σωστό και χάσατε την πρώτη μάχη ήδη του πακέτου των αποβλήτων. Χάσατε τη μάχη στην Κομισιόν. Δεν θα σας ρωτήσω λοιπόν για αυτή τη μάχη, καλύτερα να κοιτάξουμε το μέλλον και την επόμενη μάχη η οποία για μένα είναι να γίνει η αιφόρο ανάπτυξη βασικό τμήμα της ε, αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης και να εγγυηθείτε πως θα γίνει κάτι με το επενδυτικό σχέδιο του Juncker. Όλοι ξέρουμε πως η οικονομία του αύριο θα είναι μια αϊφόρος οικονομία. Οπότε αν αρχίσουμε να επενδύουμε στην αυριανή οικονομία, οι επενδύσεις αυτές ε, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια αϊφορίας. και γνωρίζουμε πως οποιαδήποτε επένδυση στην αντίθετη κατεύθυνση είναι πεταμένα λεφτά. Έχω λοιπόν τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Συζητάτε ήδη με τους συναδέλφους σας Κατάινεν και Τίμερμανς για το πώς θα διφλέξετε τα κριτήρια βιωσιμότητας και εφορίας στο σχέδιο Juncker και δεύτερον έχετε κάνει μια δική σας ανάλυση του επενδυτικού αυτού σχεδίου και του βαθμού αηφορίας και εάν ναι μπορείτε να στείλετε αυτή την ανάλυση στο Κοινοβούλιο. Εάν όχι σκοπεύετε να κάνετε μια τέτοια ανάλυση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Εγώ κοιτώντα ε, τα έργα τα οποία κυκλοφορούν από ό,τι φαίνεται για το επενδυτικό σχέδιο είναι παλαιού τύπου υποδομές ε, μεταφορών και όχι αυτό το οποίο θα λέγαμε η οικονομία και φοβάμαι πως θα έχουμε κάποιο είδους fast track για να παραμερίσουμε τις οικολογικές ανησυχίες. Μπορείτε να συμφωνήσετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και πως αντιθέτως το επενδυτικό σχέδιο του Juncker θα είναι το πρώτο βήμα προς μια αηφόρο ευρωπαϊκή οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα για την ΚΟΕ κυρία Κονέτσνα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μας δώσατε κάποιες ε, λεπτομέρειες, κάποιους ε, τομείς και πρέπει να πω πως στην ΚΟΕ δεν είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με το ότι εδώ και πέντε χρόνια προετοιμάζαμε ένα πακέτο αποβλήτων, μας απασχόλησε πολύ, κάναμε πολλές αναλύσεις και να λέμε σήμερα πως ε, θα φέρετε κάτι σε ένα χρόνο ε, δεν είναι και πολύ ικανοποιητικό αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα και ελπίζω πως με τη δική μας την ε, στήριξη και όσων ελπίζουν ότι θα πάρετε το θέμα αυτό σοβαρά θα είμαστε ε, επιτυχημένοι. Έχω κάποια ερώτηση. Είπατε πως δεν πρέπει πλέον να επιλέγουμε μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος γιατί αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Σε ποιο βαθμό είστε σίγουρος ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των δύο στην TTIP σε περίπτωση που εγκριθεί αυτή. Δεύτερον, συμφωνείτε πλέον και με τις προτάσεις της ε, Κομισιόν και μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα αποσυρθούν. Μιλάω για τις προτάσεις των τομέα αυτών. Και τέλος ε, ένα άλλο θέμα. Με, για την εφαρμογή των υφιστάμενων ε, διατάξεων για την ποιότητα του αέρα. κάτι πρέπει να γίνει για να εφαρμοστούν οι οδηγίες οι οποίες θεωρητικά ισχύουν αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να αναγκαστούν να τις ε, εφαρμόσουν γιατί όποιος δεν θέλει να τις εφαρμόσει απλά δεν τις εφαρμόζει. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την αρχική σας δήλωση πρέπει να σας πω πως ε, ε, είμαστε ευγενικοί μαζί σας μέχρι στιγμής. Εγώ ως Ολλανδός θα είμαι κάπως πιο όμως. Να σας πω τι σκέφτονται εδώ πέρα οι συνάδελφοι. Σκέφτονται πως η Επιτροπή μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για το περιβάλλον και ε, στο εσωτερικό της Κομισιόν έχει αποτύχει και πραγματικά εδώ πέρα παραβιάζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης γιατί εάν πραγματικά λέμε πως ε, θέμε να ακούσουμε πρώτα την άποψη των θεσμικών οργάνων για το πακέτο των αποβλήτων. Μα αν όλοι οι υπουργοί το Δεκέμβριο λένε πως δεν το θέλουμε και εάν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατά της απόσυρσης και αν και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων λένε στην Κομισιόν πως είναι κατά της απόσυρσης και εσείς συνεχίζετε με την απόσυρση και μετά μας λέτε πως ακούτε τα άλλα θεσμικά όργανα, ε, αυτά είναι μπουρδες. Και ε, παραβιάζετε οποιαδήποτε εμπιστοσύνη θα α, σας είχαμε. Εσείς είστε ο υπεύθυνο και πρέπει να απαντήσετε. Γιατί συνεχίζετε ενώ όλα τα θεσμικά όργανα λένε πως είναι εναντίον. Πρέπει να απαντήσετε. Και μετά, αν είναι να περάσουμε στην ουσία, να είμαι σαφής γιατί εσείς δεν ήσασταν. Λέτε πως έχουμε κάποιο όραμα για τους στόχους ε, ανακύκλωσης. Δεν είναι σαφές αυτό. Θα διατηρήσετε τους στόχους στην ομοθετική πρόταση. Ναι ή όχι. Το όραμα δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι νομοθετικές προτάσεις και θέλω στόχους εκεί. Όταν λέτε πως θα είμαστε πιο φιλόδοξοι με το να κλείσει ο κύκλος και μετά μιλάτε μόνο για έναν οδικό χάρτη, αυτό σημαίνει πως η μεγαλύτερη φιλοδοξία είναι απλά μπλα μπλα άλλη μια ανακοίνωση της Κομισιόν. Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε πως η μεγαλύτερη φιλοδοξία σημαίνει νομοθετικές προτάσεις για ολόκληρο τον κύκλο και όχι μόνο ένας οδικός χάρτης. Μόνο αν μας υποσχεθείτε αυτά τα πράγματα εδώ και τώρα μπορεί να ανακτηθεί κάποια εμπιστοσύνη γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ε, εγώ θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να τα πάρετε πολύ στα σοβαρά αυτά που σας λέω. Ευχαριστώ. Τέλος για την ευθυντή ο κύριος Μπετιτσίνη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πίτροπε. Εγώ άκουσα τα όσα μα είπατε, κυρίω όταν μιλήσατε για κυκλική οικονομία. Συνήθως όταν γίνεται λόγος για κυκλική οικονομία γίνεται, ε, γίνεται πάντα λόγος ε, από το, την πλευρά των αποβλήτων, δηλαδή καλύτερα να πάρουμε μέτρα ώστε να χρησιμοποιούνται τα απόβλητα. Ωστόσο δεν γίνεται λόγος ε, για το κομμάτι που είναι πριν, δηλαδή το να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις βασικές πηγές που χρησιμοποιούνται, τις πηγές κυρίως όταν αυτές είναι ορυκτές, τους, τους δηλαδή. Εσείς είστε όμως και για το περιβάλλον και για την αυτιλία και για την αλία. Εδώ θέλω να μιλήσω για την Κροατία και το πετρέλαιο. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση της Κροατίας έκλεισε στις 3 Νοεμβρίου το πρώτο διαγωνισμό όπου έδωσε, ανέθεσε 10 άδειε για εκμετάλλευση ε, εξορίξεων πετρελαίου που συμπεριλαμβάνουν χιλιάδες μίλια ανάμεσα στο Μαυροβούνιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, 7 χώρες, μισή Αδριατική θάλασσα δηλαδή που ανέκαθεν αποτελούσε μια πηγή πλούτου για τον τουρισμό αλλά και για την αλληλεία 4.000 ε, μίλια ακτές ε, για τα 1.300 νησιά όπου κατοικούν πολλοί άνθρωποι. Εξηγήσατε εσείς τους Κροάτες ότι με τις εξέδρες εξόριξης πετρελαίου ε, για πάντα αυτό το αλλιευτικό, ο πλούτος και ο, ο τουριστικός πλούτος της περιοχής. Το εξηγήσατε στους Ιταλούς, στους Σλοβαίνους, στους ε, Μαυροβούνιους, στους Έλληνες ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι, με τις πλατφόρμες αυτές θα υπάρξει μόλυνση για πάντα. Και όλη αυτή η κληρονομιά θα χαθεί για πάντα. Και εγώ λέω και επειδή περιμένω ότι θα μου πείτε ότι εμεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε εμεί για το ενεργειακό μείγμα τα κάτι μέλη θα το αποφασίσουν αυτό. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει ποιος θα το αποφασίσει το ενεργειακό μείγμα. Θέλω να ξέρω τι κάνει η Κομισιόν, εσείς δηλαδή, για να ε, αποφύγετε ώστε να διατηρηθούν δύο βασικά ε, θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία περιγράφονται και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή δικαιώμα στην υγεία και δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος. Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε αυτά τα δυο. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στο πρώτο σύνολο ερωτήσεων σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα 6-7 λεπτά γιατί έχουμε και άλλους που θέλουν να σας ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κατανοώ τις ε, ανησυχίες σας. Μιλάτε για απόβλητα σε επίπεδο πρώτων υλών. Ναι, ε, εκεί πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και ξεκίνησα από το τέλος αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα παράδειγμα για το πόσο πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από την παρούσα πρόταση. Τα κράτη-μέλη έχουν ασφαλώς το δικαίωμα να αποφασίσουν αν θα κάνουν εξορίξεις. Θα πρέπει όμως να σέβονται την νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Και υπάρχει στάμε νομοθεσία. Μετά, Ευχαριστώ τον Πας για την εθάρισή του. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξή. Αν ορισμένοι από εσάς είστε ικανοποιημένοι με μισό κύκλο, τι να πω, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο. Κάποιοι θέλουν να εστιάσουμε μόνο στο τέλος του δρόμου, στην κατανάλωση και στα απόβλητα. Όχι, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτή την προσέγγιση. Δεν είμαι αρκετά ικανοποιημένο. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι μόνο στην νομοθεσία. Όχι, εγώ θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος και στην εφαρμογή. Η επιτυχία μας δεν θα μετρηθεί με τον αριθμό των νομοθετικών κειμένων που θα υποβάλουμε, αλλά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Σα Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη ε, που μου υπόσχεστε. Σε ό,τι φορά την οικονομική ανάπτυξη που ε, πάει χέρι-χέρι με το περιβάλλον. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Αν έχουμε ε, πια ποια καλύτερη απόδειξη γι' αυτό από την κυκλική οικονομία. Έχουμε μία λύση, κυκλική οικονομία, η οποία λύνει και το οικονομικό θέμα, γιατί θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των πόρων, θέλουμε η βιομηχανία μας να είναι πιο ανταγωνιστική και λύνει ταυτόχρονα και το περιβαλλοντικό, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, το, της έλλειψης φυσικών πόρων κλπ. Οπότε, πράγματι συμφωνώ ότι περιβάλλον και οικονομία θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και ό,τι τον κύριο Λαμπράντη. Γκερμπράντη, συγγνώμη, λέει ο Δεν θα έλεγα ότι είχα, έχασα την πρώτη μα μάχη. Αν θυμάστε, κέρδισα την πρώτη μου μάχη με τι πλαστικέ σακούλε. Και πρέπει να υποβάλουμε μια, ένα πακέτο κοινωνικής πιο φιλόδοξο που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα απόβλητα αλλά και την παραγωγή. Και μόνο έτσι θα έχουμε κερδίσει από κοινού τη δεύτερη μάχη. Σε ό,τι αφορά με το, τη συζήτηση για το θέμα του προγράμματος στρατηγικών επενδύσεων. Είναι κάτι το οποίο συζητούμε συνεχώς. Και μάλιστα εμείς υποβάλαμε και γραπτός την ανησυχία μας. Διότι αυτά τα, τα, αυτά τα ποσά, αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να οδηγηθούν σε βιώσιμα έργα. Και θα μεριμνήσουμε ώστε αυτό να γίνει. Κύριε Γκέρλινγκ, για το πακέτο ε, ποιότητας του αέρα δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή. Προφανώς Εργαζόμαστε όμως και σε αυτό το θέμα. Αναφέρατε το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και θέλω να ξαναπώ ότι ναι, αυτό είναι ο γνώμονάς μας, αυτή είναι η βασική μας στόχη. Ματίας, δεν συμφωνείτε με την απόσυρση. Αν μιλούσαμε μόνο για την απόσυρση θα έλεγα και εγώ το ίδιο. Αλλά μιλάμε για μια απόσυρση της πρότασης που δεν σταματάει εκεί. Αν, μιλού, αν μιλούσα μόνο για μια απλή στεχνή απόσυρση θα ήμουν εξοργισμένος όπως και εσείς. Δεν μιλάμε για μια απόσυρση. Μιλάμε για μια απόσυρση προκειμένου να επανέλθουμε με μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Και για την πλευρά των αποβλήτων και για την πλευρά της παραγωγής που είναι κάτι καινούριο. Οπότε μην μπαίνετε μόνο τη μισή πραγματικότητα. Αποσύρουμε για να επανυποβάλλουμε. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και το ότι χάνουμε χρόνο. Συμφωνώ μαζί σας ότι ε, όλα πλέον συνδέονται και με την οικονομία. Οπότε ε, θα πρέπει όλες μας οι προτάσεις να συνάδουν με τους στόχους περί ανάπτυξης, ε, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Δεν χρειάζεται να χάσουμε άλλο χρόνο και αυτή είναι και η δική μου έκκληση. Αυτό που λέω είναι ας κοιτάξουμε μπροστά, ας εστιάσουμε στην καινούρια πρόταση. Γιατί λέτε χάνουμε χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε καθυστερημένοι. Και παρόλο που δεν θέλω να το πω, μερικές φορές αισθάνομαι ότι ε, αυτά που έχουμε υποβάλει ως προτάσεις είναι λίγα και καθυστερημένα. Οι συζητήσεις για τις έννοιες αυτών που παρουσιάζουμε σήμερα ξεκίνησαν τη του και πήρε όλα αυτά τα χρόνια, όλε αυτέ τι δεκαετίες για να κατασχίσουμε να τα συζητάμε αυτά συγκεκριμένα και απτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η καθυστέρηση. Όχι οι κάποιοι λίγοι μήνε που θα χρειαστούμε για να βελτιώσουμε αυτό που ήδη είχαμε προτείνει. Ματίας ξανά μίλησε για το θέμα της χρηματοδότησης. Και εγώ συζητώ με τους συναδέλφους μου Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην φάση της εφαρμογής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εστιάσουμε στην νομοθεσία να την κάνουμε πιο φιλόδοξη. Όχι. Θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος και όλη η Κομισιόν θέλει να είναι πιο φιλόδοξη στα αποτελέσματα. Με συνάδελφο Ακρέτου προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να διοχετεύσουμε περισσότερα κονδύλια σε σχέδια που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη, σε ορισμένα κράτη-μέλη, να ε, ε, τηρήσουν τους στόχους. Γιατί να χρηματοδοτούμε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στα κράτη-μέλη, ενώ θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε στη θέση τους ε, δράσεις που θα βοηθήσουν στη συμμόρφωση με την νομοθεσία. αφορά τον κύριο Μπέλετ. Για την γραφειοκρατία κλπ. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και λέμε συνεχώς, θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Όχι μέσω χαμηλώματος του πύχη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει εκθέσεις κάθε εβδομάδα, εκατομμύρια τόνους χαρτιού κλπ. το, αν μπορούσαμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό ε, των συνεχών αναφορών και εκθέσεων χωρίς να μειώσουμε τις, τα, τη, χαλαρώσουμε τους όρους τότε αυτό θα ήταν το καλύτερο. Θα επιστρέψω αργότερα να δω και κάποια σχόλια στα οποία δεν απάντησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ε, έθεσα δύο πολύ απλές και συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, και δεν έλαβα απαντήσεις. Αν έτσι θέλετε να συνεχίσουμε, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Ε, Στόχοι ανακύκλωσης θα παραμένουν στην πρόταση και δεύτερον θα υπάρξει νομοθετική πρόταση από την πλευρά της παραγωγής. Δηλαδή περισσότερη φιλοδοξία σημαίνει περισσότερες νομοθετικές προτάσεις στην πλευρά της παραγωγής. Δύο απλές ερωτήσεις με δύο απλές απαντήσεις. Μπορώ να το ζητήσω αυτό. Ναι οι στόχοι θα παραμείνουν στην πρώτη σας ερώτηση και για όσον αφορά την παραγωγή και την πλευρά της παραγωγής και την νομοθεσία περί παραγωγής και πώς θα το χειριστούμε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε γιατί θα μπορούσε να είναι ένα μείγμα νομοθεσίας ανακοινωθέντων και ε, ανακοινώσεων. Δεν το ξέρω και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Δεύτερος γύρος, 27 έχετε ζητήσει το λόγο. Και έπειτα πρέπει όλοι να μείνετε στο ένα λεπτό. Πέτερλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, χάρηκα που τονίσατε την καινοτομία και τη στρατηγική προσέγγιση και θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένος ε, ως προς αυτό. Εγώ πιστεύω πως χρειάζεται νεολογική ε, καινοτομία και διατομιακή προσέγγιση. Νομίζω πως ε, τα αγροκτήματα, κυρίως οι μικρές παραγωγικές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υποφέρουν από χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλά έσοδα. Πέρα από τα λιπάσματα και η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό πάγιο κόστος για τους γεωργούς και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε στην παραγωγικότητα του γεωργού. Ένας ε, Γεωργός μέσω εγγυημένων ενεργειακών τιμών θα μπορούσε να εγκαταστήσει ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας που θα χρηματοδοτείται μέσω μιας γραμμής πίστοσης. Ένα κομμάτι της ενέργειας θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί ο, Γεωργό, ο ο Γιώργος και το υπόλοιπο να δίνεται σε ένα FES ε, πλέγμα. Έτσι θα πρέπει να είναι εγγυημένη η τιμή της ε, κιλοβατόρας. Ε, έτσι θα μπορούσε και ο Γιώργος να έχει ένα επιπλέον εισόδημα και να εξασφαλίζει τις ανάγκες του σε ενέργεια. Μου είπατε ένα λεπτό, γι' αυτό διάζομαι. Αυτό που χρειάζεται είναι να ολοκληρωθούν οι τηλεπικοι... επίσης οι τηλεπικοινωνίες. Το ερώτημά μου είναι πώς θα μπορέσετε να στηρίξετε ένα τέτοιο συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ. Dear colleagues, uh, we have to... Συνάδελφοι, πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας, γιατί ξέρετε, έχουμε χρονικούς περιορισμούς. Και Γι' αυτό σας καλώ να κρατήσετε αυτό το χρονικό όριο του ενός λεπτού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής κύριε Επίτροπη γιατί αναφέρετε ότι το 2015 είναι ε, ε, ένα έτος ε, για το περιβάλλον αλλά και επίσης επειδή είπατε ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά την εφαρμογή. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις για την εφαρμογή αλλά και τη βιοποικιλομορφία πώς θα ε, εφαρμόσετε τα μέτρα που προβλέπονται για τα ε, είδη τα οποία ε, μπαίνουν μέσα στα οικοσυστήματα, τα επιθετικά είδη και έπειτα θέλουμε, ε, μάλλον δεν υπάρχει εξαίρεση στην οδηγία περί αποδημητικών πουλιών ε, για τα πουλιά που περνούν πάνω από τη Μάλτα. Εσείς τι κάνετε για την προστασία αυτών των ειδών που είναι υπό εξαφάνιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βυσνιεύσκα. συζητήσαμε μόλις για την οδηγία περί μονάδων, μεσαίων μονάδων καύσης. Πιστεύω πως οι οριακές τιμές που προτείνει η Κομισιόν θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Ο κόσμος δηλαδή θα απομακρυνθεί από την κεντρική θέρμανση και θα αγοράσει ο καθένας δικό του καυστήρα και θα καίει ό,τι να είναι. Ε, ακόμα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να καίγονται εκεί μέσα. Να τονίσω επίσης το γεγονός ε, του ενεργειακού αποκλεισμού, ένα φαινόμενο που αυξάνεται στην Ευρώπη. 1,5 εκατομμύριο Πολωνοί απειλούνται από την ενεργειακή φτώχεια αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν καν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Θα μπορούσαμε εύκολα να φτάσουμε στα 150 εκατομμύρια κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν μια ρεαλιστική πολιτική που θα εγγυάται την πρόσβαση στην θέρμανση και στην ενέργεια για τον κόσμο που αντιμετωπίζει δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Παρακαλώ την Κομισιόν λοιπόν αυτό να το λάβει υπόψη. Είμαι ευτυχή που ο να θα αναθεωρήσει την πρότασή του, αλλά θα ήθελα να είναι πιο ευέλικτο στην χρήση ε, άνθρακα. Ακόμα και αν είναι λίγο χειρότερο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ε, συνθήκες. Θέλουμε όμως να χρησιμοποιήσουμε το, όλο το δυναμικό της κεντρικής θέρμανσης και της συνπαραγωγής. Ευχαριστώ κυρία ε, ε, ε, Πέρυσι υποστήριξε το Beater, συγγνώμη, υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταπολέμηση της των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και είπατε ότι θα δουλέψετε για να χειριστείτε το θέμα, αλλά δεν δεσμευθήκατε για ένα πρόγραμμα δράσης. Έχετε πολλά να κάνετε με την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα πτηνά και το, το, ε, το habitat των, ε, των πουλιών έχετε πολλά να κάνετε, ωστόσο παραμένει αυτό κομμάτι της δουλειάς σας. Εγώ θέλω να εστιάσω ε, σε αυτό όμως το θέμα. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι πρόοδο έχετε σημειώσει όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής. Θα προτείνετε κάποιο πρόγραμμα δράσης σε σύντομα και πότε αναμένετε να ολοκληρώσετε την εξέταση του 7ου προγράμματος ε, και των μέτρων σκοπιμότητας όσον αφορά την ε, αποψήλωση των δασών. Τέλος, τι σκοπεύετε να κάνετε μετά από την επίσημη σημείωση προς τη Μάλτα ε, όσον αφορά την ε, παγίδευση του, της καρδερίνας. Ο κύριος Αμαριέ. Ε, ευχαριστώ. Η ερώτησή μου θα είναι σύντομη. Η Κομισιόν αποφάσισε να διοργανώσει την εξαίρεση της οδηγίας για τους οικοτόπους των πτηνών της, της εδά τα υπερπόντια εδάφη και τα εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό είναι μυστήριο διότι εκεί, εκεί μένουν τα περισσότερα ε, πτηνά που είναι υποκίνδυνο. Ε, ρώτησα γραπτό στην Κομισιόν και μου απήντησαν ότι δεν ε, προτίθεται και δεν σκοπεύουν, δεν σκέφτονται μάλλον να αναθεωρήσουν την οδηγία τους για να συμπεριλάβουν και τα απομακρυσμένες περιοχές. Σε πραγματικά έχω μείνει ξερός. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι περιοχές σε αυτή την ε, οδηγία, θα, μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης θα εξετάσετε αυτό το θέμα όπως ελπίζω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σλέκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σήμερα ακούσαμε ε, ένα νέο ορισμό των λέξεων απόσυρση και φιλόδοξη στόχη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν ανάντι στην κυκλική οικονομία για να έχουμε περισσότερη χρήση, περισσότερη ανακύκλωση, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Καμία νομοθετική δράση φέτος για κανένα ε, τέτοιο μέτρο το πολύ πολύ μία ανακοίνωση ανταυτού. Θα δούμε ένα τροποποιημένο πακέτο περί αποβλήτων, νέους στόχους ε, επίσης ε, και νέα αύξηση της, της αποτέφρωσης ανακυκλωμένων και μη ανακυκλωμένων αποβλήτων. Και περνάμε έτσι στο έβδομο πρόγραμμα δράσης το οποίο ε, αντιθέτως ζητάει και πάυση της ε, ταφής ε, και μείωση της αποτέφρωσης. Ίσως όμως μία λύση για το πρόβλημα της ενεργειακής ένεσης θα μπορούσε να είναι η αποτέφρωση για να παράγει την ενέργεια. Το ερώτημά μου είναι η πρόταση, η πιο φιλόδοξη που θα δούμε είναι καμία νομοθεσία, μικρότερη αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και λίγο και ναι, δεν θα κάνετε τίποτα για, την, ε, για τις ε, χωματερές και την αποτέφρωση. Σας ευχαριστώ, Έντι. Sì, grazie Presidente, buongiorno Commissario. Η συνάδελφος Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και Επίτροπε. Εγώ μόλι ολοκλήρωσα το σχέδιο γνωμοδότηση όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων, πράσινων θέσεων απασχόληση και δούλεψα με βάση την ανακοίνωση τη Επιτροπή. Είχα την εντύπωση πω αυτή η νέα Κομισιόν καταρχήν δεν ε, βρίσκει πια τι να κάνει ανάμεσα στι διάφορε πρωτοβουλίε που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόληση και αναφέρομαι για παράδειγμα στην απόσυρση τη πρόταση αναθεώρηση τη οδηγία για την απόβληση που θα κοστίσει 180.000 πράσινες θέσεις απασχόλησης. Εν γέννη έχω την εντύπωση πως αυτή η Κομισιόν δεν σκοπεύει να δώσει συνέχεια σε εκείνη την πολιτική στάση που θα ξεπερνούσε την οικονομική κρίση βασιζόμενη στην πράσινη οικονομία. Μάλιστα φαίνεται να έχει στερηθεί κάθε περιεχομένο αυτή η ερώτηση. Το ερώτημά μου αφορά, μάλλον είναι πέρα από τα απόβλητα των τον ε, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσετε, ποια μέτρα θα θεσπίσετε για να κινητοποιήσετε την πράσινη οικονομία και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης όπως, απασχόλησης, όπως έχει αναφέρει η Κοικομισιόν τα περασμένα χρόνια. Σας ευχαριστώ και τώρα ο συνάδελφος ε, Πάλτσο. Ε, σας ευχαριστώ. Βλέπουμε το βλέπουμε πως έχουμε ένα έτος ε, φυσικών ε, πόρων, οι οποίοι οπωσδήποτε παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά συχνά τα δάση που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πόρος τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως βιομάζα. Αν συνεχίσουμε έτσι θα κινδυνεύσουν τα δάση και η βασική τους ε, λειτουργία. Μία απλή ερώτηση για εσάς. Θα ήθελα να επαναλάβω την ερώτηση του κυρίου Άικχαουτ και θέλω συγκεκριμένη απάντηση από εσάς. Γιατί αποσύρθηκε το πακέτο διαχείρισης αποβλήτων. Μας λέτε πως θέλατε να καταθέσετε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Ποια είναι η φιλοδοξία λοιπόν. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο, όχι οράματα. Ευχαριστώ κύριος Γκάμπους. Επίτροπε, σε ό,τι αφορά την απόσυρση του πακέτου για την κυκλική οικονομία, να σας πω ότι εμένα μου αρέσει να κοιτάω προς το μέλλον και ελπίζω η πρόταση που θα υποβάλλετε να είναι πράγματι φιλόδοξη. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις όμως έχω να σας κάνω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το σαλιγκάρι του Δέλτα του Εύρου. Το 2012 ε, είχατε πάρει μια απόφαση η οποία ε, παρατάθηκε. Πιστεύετε ότι αρκεί για να ε, λύσει το πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή εντοπισμένο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης. Τα σαλιγκάρια δεν εξαφανίστηκαν τα δύο τελευταία χρόνια και αυτό αποτελεί σημαντικό κίνδυνο να επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, τι μέτρα θα πάρετε για να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα της Μεσογείου στην κοινή αλευτική πολιτική σε ένα θέμα όπως η υποχρέωση ε, της εκφόρτωσης ε, μεγεθών που είναι αντικανονικά. Που αυτή την ε, στιγμή αυτά τα μικρά μεγέθη ρίχνονται στη θάλασσα και αυτό βοηθάει τον, τον πληθυσμό των ηχθείων στη θάλασσα. Τι θα γίνει τώρα. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντάνς. Πολύ καλή προσήλωσή σας για τη μειώσιμη ανάπτυξη. Και ένας από τους πυλώνες της είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητήσει με άλλους εταίρους τους ε, στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας, μία από τις περιοχές ε, τις οποίες θέλει η Κομισιό να είναι ε, δραστήρια. Τι θα κάνετε για να μας καθησυχάσετε ότι όταν συζητηθεί η ατζέντα του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κατηγορηθεί για ε, διπροσωπεία όταν μιλάμε τους εταίρους μας. Δεδομένου ότι αποσύρεται το πακέτο για τα απόβλητα. Κύριε Ντάνκαν. Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες πουλιών και οικοσυστημάτων και το refit, πολλά έχουν ξεκινήσει ή έχουν αλλάξει από όταν υποβλήθηκαν αυτές τις προτάσεις. Για παράδειγμα στην Σκοτία έχουμε σύγκριση αυτή τη στιγμή ε, μεταξύ των πάρκων ανεμογεννητριών και των φύλων των πτηνών. Έχουμε την οδηγία περιχωταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα, ε, αλλά πώς θα χρησιμοποιηθεί. Στη Βόρεια Θάλασσα έχουμε πολλές δραστηριότητες που δεν υπήρχαν παλιότερα. Για παράδειγμα, ανανεώσιμες ε, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μετακινούνται όλο και πιο μέσα στη θάλασσα έχουμε παραδοσιακού χρήστε κλπ. κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Ερώτηση είναι πώ θα λειτουργήσει αυτό το εργαλείο του χωροταξικού σχεδιασμού. βράχει πρόθεσμα. Thank you very much. And now Mr. Olveni. Ο κύριος Olveni. The chairman, uh, very briefly on my Σα ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή υπόσχεται μια έκθεση ε, νομοθεσία για τα απόβλητα των ορχείων. Στην έκθεση αυτή θα ληφθούν υπόψη οι αδυναμίες που υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων για τα ε, ορυχεία. Θα ληφθούν μέτρα, νομικά και άλλα, για την ε, εφαρμογή των κανόνων. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, διότι ε, είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό σημείο αφετηρίας. Μιλήσατε για διμερείς, συμφων... συζητήσεις πράγματι και εγώ σε επισκέφθηκα την περασμένη εβδομάδα για να μιλήσουμε για την καταστροφή στο ΤΙΣΑ πριν από 15 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για τέτοια θέματα. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία. Ε, κοιτάξτε, συγκεκριμένα να σας πω το εξής. Ε, συχνά Αναφερθήκατε στην οδηγία για τους βιοτόπους και τα πτηνά και το ερώτημα είναι πως από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη αμελούν τις υποχρεώσεις τους ε, εδώ πέρα και θα πρέπει νομίζω να γίνει κάτι και στο πλαίσιο του fitness check της ε, βιομηχανίας γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα επιβλέπουμε τόσο έντονα την εφαρμογή αυτής της νομοσίας και θα καταλήξουμε σε μια πλημελή εφαρμογή της. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε πως θα έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας χωρίς επιδείνωση της ε, προστασίας. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, για το χρηματοδοτικό μέσο φυσικού κεφαλαίου. Είπατε πως θα προωθηθεί και η βιοπικιλότητα. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε πως ένα κομμάτι αυτών των 120 εκατομμυρίων ευρώ θα πάει και σε έργα βιοπικιλότητας. Έχετε κάτι συγκεκριμένο κατά νου. Ευχαριστώ. Κύριε Σφαγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είχα διάφορες αμφιβολίες. Εδώ, εδώ είμαι, κύριε Επίτροπε. Εδώ κάθομαι. Εδώ, εδώ, στο, στη μέση. Είχα διάφορες ερωτήσεις ε, να κάνω, αλλά θα κάνω μία για τη θάλασσα και την αλία. Θεωρείτε ότι ε, συνοθή, μάλλον συναντηθήκατε με την Υπουργό μας ε, στις 16 Φεβρουαρίου. Ένα από τα θέματα ήταν η αλία του Καρχαρία της Μαδέρα. Ε, η κυρία Υπουργό σα ανέφερε τα παράπονα των αλληλευτικών κοινοτήτων της Μαδέρας ε, και των Αζωρών σε σχέση με την τυχαία ε, αλληλεία αυτού του είδους. Ωστόσο αυτή απαγορεύεται. Έχει σταλεί και γραπτή ερώτηση ε, στην Κομισιόν ε, για αυτό το θέμα. Εσείς πιστεύετε πως ε, αυτή η ε, αποτελεί κίνδυνο και γι' αυτό το είδος και ότι θα πρέπει να προστατευτεί αυτό το είδος που κινδυνεύει από εξαφάνιση. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε σχετικά μήπως θα μπορούσε να ακυρωθεί ο εν λόγω κανονισμός ώστε αυτού του είδους η τυχαία αλληλεία να μην γίνεται πια. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και άλλοι συναδελφοί θα ήθελα και εγώ να αφαιρθώ στο θέμα της Natura 2000 ε, των βιοτόπων και των πτηνών μιλήσατε για έναν επανέλεγχο που θα γίνει. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που βλέπετε και να μας πείτε εάν βλέπετε μία ανάγκη μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν θεωρείτε πως έχουμε πρόβλημα εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Εμείς ε, βλέπουμε στη χώρα μου πως ε, έχουμε μία μετατόπιση θα έλεγα των, της σχετικής ε, νομοθεσίας. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η αρχική πρόθεση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριος Λάγκεν. Αναφέρατε το 7ο πρόγραμμα δράσης και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 και εδώ πέρα ξεκινάμε με την περίφημη πολιτική οικολογικών προϊόντων ε, και το ερώτημα είναι τι σκοπεύετε να κάνετε για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Άκουσα και τον αντιπρόεδρο Τίμερμανς που λέει πως δεν χρειάζεται κάθε πρόβλημα ένα νόμο. Αυτό ίσως, αλλά όταν μιλάμε για την πολιτική των προϊόντων χρειάζονται προδιαγραφές που θα ισχύουν για όλους. Και αυτό δεν γίνεται με εθελοντικά μέτρα χρειαζόμαστε νόμους ε, με δεσμευτικές προδιαγραφές. Δεύτερο ερώτημα, πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Νομίζω θα βοηθούσε διάφορες ενώσεις να έχουν πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Τι άποψη έχει αυτό. 60 δευτερόλεπτα ακριβώς. Σας ευχαριστώ, Ντέμες Μακερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, ως και ο δισηγητής της ομάδας μου για την κυκλική οικονομία. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση για το πρόγραμμα του 2015. Προσπαθούμε βεβαίω να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, αλλά έχουμε κάποια επιφυλακτικότητα. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Τι εννοείται ακριβώς όταν λέτε πώς θα γίνει ο φάκελος πιο προσαρμοσμένος στις χώρες. Μετά μιλήσατε για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Πώς συμβιβάζεται αυτό με αυτό το οποίο μας είπατε για περισσότερη φιλοδοξία όσον αφορά την εφαρμογή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ίσως μια επικοδομητική συνεισφορά υπάρχει η μοναδική δυνατότητα που, έχει τώρα, που έχετε με την έκθεση της φωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Τέλος, η περιφέρειά μου, η Φλάνδρα, έχει κάποιες ε, πρωτοποριακές ιδέες ε, και πρωτοπόρους στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Οργανώνω μια σχετική εκδρομή λοιπόν και ελπίζω να είστε παρόν. Ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίαση των σχεδίων σας θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 3.000 περιπτώσεις που ο κόσμος άρρωσταίνει λόγω μικροβίων τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Στη δε Γερμανία από ό,τι φαίνεται 700 χιτώνει αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην γεωργία. Δηλαδή πάνω από τα διπλάσια από ό,τι στα ανθρώπινα και από ό,τι φαίνεται σχεδόν όλο το κρέας γαλοπούλας ε, έχει αντιβιωτικά. Θα ήθελα λοιπόν να μας τι κάνει η Κομισιόν για αυτές εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις. Πρώτον προβλέπονται κάποια μέτρα για την περιορισμό της χρήσης αντιβιωτικών στη γεωργία ακόμη περισσότερο. Δεύτερον, προβλέπονται κάποια μέτρα έτσι ώστε να μην φτάνει κρέας ή προϊόντα κρέατος που αποδεδειγμένα ε, είναι μολυσμένα με μικρόβια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα αντιβιωτικά να μην φτάνουν αυτά στο εμπόριο. Ευχαριστώ κυρία Ριβασί. Δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτον, ε, σε ό,τι αφορά την διάλυση των σκαφών. Όπως γνωρίζετε όλο και περισσότερα σκάφη στο τέλος ζωής τους ε, διαλύονται συνήθως στην Ασία σε πολύ άσχημες συνθήκες τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον όσο και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους. Το 2013 υιοθετήσαμε μια οδηγία και μπορεί μάλιστα να επιταχυνθεί η εφαρμογή της ε, όταν η Κομισιόν ε, δημοσιεύσει τον κατάλογο των χωρών οι οποίες μπορούν να διαλύουν με οικολογικό τρόπο αυτά τα σκάφη. Ερώτηση λοιπόν, ε, θα δημοσιευθεί αυτός ο ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνεται αυτό στο πρόγραμμα της τη Κομισιόν. Τώρα, με τον άλλο μου ρόλο, σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, υπάρχει η σύμβαση τη Μίνα Μάτα, ε, πού βρίσκεται το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής τόσο για την απαγόρευση των, της εξόριξης όσο και για την απαγόρευση της χρήσης ε, ε, του, της ουσίας αυτής στα στραγίσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλώ για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και το Natura 2000, δημιουργία δηλαδή ενό ε, πλαισίου θαλασσίων περιοχών μέχρι το 2020 ε, που θα είναι προστατευόμενες. Λέει ότι για την Αδριατική και το Ιόνιο θα πρέπει μέχρι το 2020 να φτάσουμε σε μια επιφάνεια 10% ε, που θα προστατεύεται. Αυτή τη στιγμή είναι 0,4% οι προστατευόμενες περιοχές. Μόνο 5 χρόνια όμως μένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Ποιες είναι οι ενέργειες που σκοπεύετε να κάνετε για να πετύχετε αυτούς τους στόχους και αν υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης ε, σχετικά με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Πέτιε. Πετήρ, με συγχωρείτε. i predstavlja stoljetnu tradiciju način rješavanja egzistencije osobito na otocima u Jadranu. Hrvatski ribari zbog posebnosti Jadrana koriste specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji, što je dovelo nažalost do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao u Teksasu. hoće parhi kapio problema tehniko. Should I start from beginning? Or? Ναι, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή γιατί δεν καταλάβαμε. Μάλιστα, τώρα διορθώθηκε το πρόβλημα. Έχουμε παραδόσεις αιώνων, ιδιαίτερα για κάποια ε, νησιά της Αδριατικής. Οι Κροατοί ε, αλληλείς χρησιμοποιούν και διαφορετικά εργαλεία. Ε, διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στην Ένωση, πράγμα το οποίο οδήγησε στην κατάργηση της μικρής βιοτεχνικής αλληλείας. Έχει λειτουργήσει αυτό ως μπούμεραγκ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από εσάς κύριε Επίτροπε τι σκοπεύετε να κάνετε ε, δεν ισχύουν οι ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις για όλους. Ε, η μικρή κλίμακα κασαλία θα πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί ως πολιτιστική κληρονομιά. Και θα ήθελα και εγώ να αντιδράσω στη δήλωση του κυρίου Πελιτσίνη που ρώτησε τον Επίτροπο να προειδοποιήσει την Κροατία έναντι της επιθανής εκμετάλλευσης πετρελαίου στην Αδριατική και τα σχετικά προβλήματα. Θα πρέπει να πω ότι προσωπικά είμαι κατά της ε, εκμετάλλευσης του πετρελαίου στην Αδριατική, αλλά η Κροατία αυτή τη στιγμή ακόμα διερευνά την υπόθεση. Αντίθετα από την Ιταλία που έχει ήδη εννέα πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου και ζήτησε άδεια για δημιουργία ακόμα 19 κύριε Βέρλα, μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή του κύριου Περλιτσίνη στους, την προσοχή του στους κινδύνους που προκαλούνται από αυτές τις πλατφόρμες εξόδου πετρελαίου. Σας ευχαριστώ όλους. Για τις ερωτήσεις σας θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για απαντήσεις. Έχουμε 7-8 λεπτά άντε 10 maximum. Thank you very much, Mr. Chairman. Ε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ε, που άγγιξαν όλες τις στοιχές της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και κατάλαβα ποιε είναι και οι προτεραιότητε. σας. βεβαίω στον χρόνο που έχουμε ε, δεν μπορώ να απαντήσω σε ε, όλα αυτά, αλλά σας διαβεβαιώ πως τα σημείωσα και εγώ και οι συναδελφοί μου. Να προσπαθήσω λοιπόν τώρα να απαντήσω σε κάποιες από αυτές. Πάρα πολλοί από εσά αναφέρατε την κυκλική οικονομία και νομίζω πως ήμουν σαφής για την κατεύθυνση στην οποία εργάζεται η Κομισιόν και είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω κινήσεις από την πλευρά σας όμως ας μην κάνουμε τώρα εικασίες ε, για το τι θα περιέχει ακριβώς η πρωτοβουλία αυτή. του μήνε που έρχονται είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις δικές σας ιδέες ε, για να δούμε πώς ακριβώς είναι αυτή η πρόταση θα ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέλετε. Συμφωνούμε πως το καλύτερο είναι να προλαμβάνουμε την δημιουργία αποβλήτων ε, στο νέο πακέτο, γι' αυτό ακριβώς αναθεωρούμε το πρώτο, πακέτο, το πρώτο μέρος του φυστάμενου πακέτου και βεβαίως ε, Καλό είναι να εγκριθεί και η δική σας η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας πριν από το καλοκαίρι. Και αναμένουμε την ολοκλήρωση της ε, εργασίας σας ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, τις άλλα ζητήματα για την Natura 2000, βιοτόπους, τα πτηνά κτλ. Και σημείωσα τις ανησυχίες σας για τον επανέλεγχο αυτής της υπόθεσης και βεβαίως ε, θα φροντίσουμε να διατηρήσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο και προδιαγραφές προστασίας. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός της ε, επανέξατησης αυτής, ε, να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας με μικρότερο διοικητικό βάρος χωρίς να μειωθούν οι γενικοί στόχοι. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, η Κομισιόν θα κάνει αυτή την αξιολόγηση με τρόπο διαφανή σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους και σημαντικό είναι βεβαίως να ακούσουμε όλες τις απόψεις και βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις απόψεις τις δικές σας για να έχουμε ένα ε, επιτυχές αποτέλεσμα. Θα επανέλθουμε δε με τα αποτελέσματα του ε, ελέγχου αυτού και της δημόσιας διαβούλευσης αρχές του επομένου έτους. Για τα πτηνά στη Μάλτα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει και στο παρελθόν θα φροντίσουμε και θα φροντίσω να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να εφαρμοστεί. Η διαδικασία, όπως ξέρετε, συνεχίζεται όσον αφορά Την οδηγία για τα πτηνά και το πώς εφαρμόζεται στην Μάλτα. Τώρα για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης συμφωνώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ανακοίνωσή μας επίσης ε, θα αναφέρει το πώς θα γίνει η εφαρμογή του εβδόμου αυτού πακέτου για αυτά τα οποία είπε ο κ. Φολβένη και για την εξορρεκτική βιομηχανία θα το συζητήσουμε διμερώς, θα το συζητήσει και με άλλους όσον αφορά τώρα κάποιες διευκρινήσεις για το πώς θα προσαρμοστούμε ανά χώρα Κοιτάξτε, γεγονός είναι πως κάθε χώρα έχει διαφορετικές καταστάσεις και έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ασθενέστερα κράτη-μέλη, πού βρίσκονται τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις για να προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους, έτσι ώστε αντί να μειώνονται οι στόχοι, να ε, υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν τους στόχους. και νομίζω πως η Κομισιόν έτσι θα είναι καλύτερη στο ρόλο της ε, να δρά δηλαδή με τρόπο που να διευκολύνει τα κράτη-μέλη και όχι μόνο ως ε, ρυθμιστής. Τώρα για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη ε, υπάρχει ήδη αυτή η πρωτοβουλία. Θέλω ό,τι κάνουμε να είναι συνεπές με τις πολιτικές δραστηριότητες της ε, Κομισιόν και με τις αρχές της καλύτερης ρύθμισης και από όταν ανέλαβα εγώ τα καθηκοντά μου οι υπηρεσίες μου είχαν μια σειρά ε, ανταλλαγών απόψεων με διάφορους ενδιαφερομένους. Ε, καθώς όμως οι, συνεχίσεις, οι συζητήσεις συνεχίζονται, δεν μπορώ να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή, είναι να σας ενημερώσω αργότερα ευχαριστώ Για την ανακύκλωση, ναι, κύριε Ριβάζη, ε, μας υποχρεώνει ο κανονισμός να, να θεωρήσουμε μέχρι του χρόνου και θα το κάνουμε και θα τηρήσουμε αυστηρά και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς αλλά και εξίσου σημαντικό και τις υπόλοιπες πτυχές. Θέλω πράγματι να σταματήσει αυτή η πρακτική να διαλύονται τα ευρωπαϊκά πλοία σε παραλίες Για τα άλλα ζητήματα που λέτε, πράγματι θα δώσω και κάποιες γραπτές απαντήσεις, ε, όπως και σε άλλα ζητήματα στα οποία δεν είχα χρόνο να απαντήσω επαρκώς. Σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Να σας πω τώρα τι θεωρώ εγώ πως δεν μας απασχόλησε, δεν αναφερθήκαμε πάρα πολύ στην ε, διακυβέρνηση των ωκεανών, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, μεγάλη μας προτεραιότητα και νομίζω πως το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχιστεί ο διάλογος στους επόμενους μήνες και Αναμένω την επόμενη ευκαιρία που θα έχω να συνομιλήσω με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φαΐε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κάνω δεύτερη φορά την ερώτηση για τους ε, καρχαρίες ε, και την αλληλεία τους. Έκανα ερώτηση κομισιών, δεν μου απαντήσατε. Γραπτή δεύτερη φορά προφορική ερώτηση δεν μου απαντάτε. Ε, και, τώρα δεν μου απαντάτε. Δεν με προσέχετε. Έπρεπε να σταματήσω. Ε, μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, μια σύντομη. Απάντηση. Μα... Μέχρι στιγμής νομίζω πως ε, Έχουμε λάβει τον ε, δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων μετά την κυρία Μογκερίνη και από όσο ξέρω απαντήσαμε σε κάθε ερώτηση. Θα το δω, θα το δω. Οπωσδήποτε θα σας απαντήσουμε ε, το στομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ ε, μια γραπτή απάντηση στην ερώτησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, λέει ο Επίτροπος. Βεβαίως. Uh, when, uh, Είναι σαφές. Πως όταν, λαμβάνει πολλές, όταν δέχεται πολλές ερωτήσεις, ο Επίτροπος δεν μπορεί να απαντήσει στο λίγο χρόνο που έχει. Γι' αυτό τον ζητάμε, του ζητάμε να απαντήσει γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις που δέχτηκε. Τελειώνουμε εδώ. Τρεις η ώρα με την ψηφοφορία.